Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε στη συνεδρίασή μας. Είναι η πρώτη φορά που η συνεδρίασή μας που συνεδριάζουμε σε αυτή την αίθουσα για αυτούς οι οποίοι ακολουθείτε, παρακολουθείτε άλλες γλώσσες. Θα έχουμε τα τουρκικά στο κανάλι παριθμών 6. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για την παρουσία της Λέιλα Σάνα βραβείο Σαχάρο 1995. Και το θέμα μας σήμερα είναι το θέμα της ελευθερίας έκφρασης και των δικαιωμάτων των γυναικών στην ε, Τουρκία, αλλά φυσικά θα ασχοληθούμε και με άλλα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Και δεν πρόκειται μονάχα για την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία έχει συγκαλέσει αυτή τη συνεδρίαση, Έχουμε μαζί μας την Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα του Φύλου με τον κύριο Γκούσταυσον, ο οποίος είναι παρόν ο πρόεδρος αυτής της Επιτροπής και επίσης μαζί με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία. Η Ελένη Φλότερ, η πρόεδρος, δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας, αλλά η Ελένα Ακοπά, που είναι αντιπρόεδρο, είναι μαζί μα. Θέλω να σα ευχαριστήσω λοιπόν για τη συμπροεδρία που παρέχεται σε αυτή τη συνεδρίαση. Είναι πολύ γνωστή η αγωνίστρια η Λέιλα Λάζανά και ανεξάρτητη βουλευτής στο τουρκικό κοινοβούλιο από το Δία Μπακέρ στην νοτιοανατολική Τουρκία το 1991. Η Λέιλα Λάζανά ήταν η πρώτη κουρδικής καταγωγής γυναίκα που εξελέγει στο τουρκικό κοινοβούλιο. Το τελευταίο τμήμα του κοινοβουλευτικού της όρκου το, το είπε στα κουρδικά και αυτό οδήγησε στην άμεση σύλληψή της. Έμεινε στη φυλακή 10 χρόνια λόγω του πολιτικού της ακτιβισμού που θεωρήθηκε από τα τουρκικά δικαστήρια ότι απειλούσε απειλή για την, ε, αποτελούσε απειλή για την ακεραιότητα της Τουρκίας. Πήρε το βραβείο Σαχάροφ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1995, αλλά μόνο το 2004 και μετά μπόρεσε να το πάρει. Επανεξελέγει στο τουρκικό Κοινοβούλιο πέρσι, το 2011, και πρόσφατα η κυρία Σανά έχει αντιμετωπίσει δικαστικές διώξεις εναντίον της και ε, καταδίκες σε φυλάκιση. Πρόσφατα καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 ετών για την κατηγορία ότι διαδίδει προπαγάνδα επί τη βάση ομιλιών που έκανε το 2007-2008 μεταξύ αυτών και μια ομιλία που έκανε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προστατεύεται προς το παρόν από την κοινοβουλευτική της ασυλία. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι ο πρόεδρος μας, ο κύριος Σούλτς, επισκέφθηκε την Τουρκία στις 11 Ιουνίου και επίσης στην έναρξη της Ολομέλειας του Στρασβούργου τον Ιούλιο ζήτησε μια δίκαια δίκη για την Λέιλα Ζανά. Παρακολουθούμε λοιπόν από τη δική μας πλευρά όσο μπορούμε καλύτερα τα τεκτενόμενα σε σχέση με αυτή την υπόθεση η Τουρκία εξακολουθεί να, είναι, ε, να έχει ενώπιον τις σημαντικές προκλήσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής μας και μέσα στα πλαίσια φυσικά και της διαδικασίας ένταξης της Τουρκίας και της ετήσιας έκθεσης προόδου. Θέλω να υπογραμμίσω εξ αρχής ορισμένες πρόσφατες περιπτώσεις που έχουμε παρακολουθήσει. Από τον Οκτώβριο ως το Δεκέμβριο του 2011 δεκάδες συγγραφέων, ακαδημαϊκών, εκδοτών και δημοσιογράφων συνελήφθησαν σαν τμήμα μιας μεγάλης αντιτρομοκρατικής εκστατείας με στόχο να ε, εξαρθρωθεί ένα υποτιθέμενο τρομοκρατικό δίκαιο. Περιλαμβάνονται ο, ο Ρατζιπ Ζαρακολού που απελευθερώθηκε στις 12, στον Απρίλιο του 2012 και περιμένει να δικαστεί και είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην ε, Τουρκία και επίσης μέλος της Ένωσης Συγγραφέων στην φυλακή. Επίσης, η καθηγήτρια Μπούρσα Εσανλή από το Πανεπιστήμιο του Μαρμαρά κατηγορείται και μπορεί να αντιμετωπίσει δίκη και που επισύρει ποινή πάνω από 20 ετών στη φυλακή. Συνάντησα την κυρία Εσράλη στην φυλακή στην Κωνσταντινούπολη σε 9 Μαρτίου και κατανόησα ότι και αυτή δεν μπορεί να προετοιμάσει πλήρω την υπεράσπισή της με το συνήγορό τη, γιατί δεν της έχουν ε, απαγγείλει ακόμα συγκεκριμένη κατηγορία. Και η κυρία Μπακτάη επίσης, η οποία είναι μεταφράστρια, ερευνήτρια και ακτιβίστρια στον τομέα τη ειρήνης. Συνολικά έχουμε 193 ακτιβιστές υποκατηγορία. Η, η δίκη τους ξεκίνησε στις 2 Ιουλίου. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν ανησυχούμε τα μάλα για αυτήν την δίκη και την ενδεχόμενη ε, αυθαίρετη εφαρμογή της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας στην Τουρκία. Θα παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη σε αυτές τις δικαστικές υποθέσεις. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ακτιβιστών και αγωνιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διανομένων και συνδικαλιστών που αντιμετωπίζουν περιορισμούς και ακόμα και ε, ποινικέ ε, κατηγορίες. Μου υπενθύμησε η κυρία Κόπα ότι ήταν και η Πινάρ Σελίκ σε μία από τις συνεδρίασεις της Μικτής Επιτροπής, μια φεμινίστρια, ε, κοινωνιολόγος, συγγραφέας και ακτιβίστρια για τα θέματα ειρήνης και ισότητας των φύλων, η οποία, πάνω από την οποία επικρέμαται μια ποινή ισοβίων δεσμών για ένα δίκημα για το οποίο όμως έχει ήδη αθωωθεί δύο φορές. Θα μπορούσα να συνεχίσω να αναφέρω τις ε, διώξεις κατά συνδικαλιστών Απλώς όμως θέλω να συνοψίσω και να πω ότι παρακολουθούμε από κοντά την μεταρρύθμιση στο δικαστικό τομέα και την διαδικασία σύνταξης ενός νέου συντάγματος στην Τουρκία. Ελπίζουμε και προσδοκούμε ότι αυτά θα φέρουν θετικές αλλαγές στην Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παροτρύνει επίσης την ε, δημιουργία μιας νέας θετικής ατζέντα για να υπάρξει νέα όθηση στην διαδικασία ένταξης και ένα από τα στοιχεία αυτής της θετικής ατζέντα είναι το θέμα της πολιτικής μεταρρύθμισης και της προάσπισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Έχουμε λοιπόν αυτό το πλαίσιο περιπτώσεων και δικαστικών υποθέσεων που παρακολουθούμε και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μιχαήλ Γούσταυσον, τον πρόεδρο της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών, για να κάνει και αυτό στην, τα εισαγωγικά του σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Λέιλα Ζανά σε αυτή τη συνεδρίαση. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που δέχτηκε την πρόσκλησή μας να παραστεί στην συνεδρίαση. Επίσης χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που κάνουμε την προσπάθεια μαζί, δηλαδή έχουμε μια κοινή συνεδρίαση. Είμαι εδώ ως πρόεδρος της δικής μου επιτροπής και έχουμε και άλλα μέλη της Επιτροπής Ότιας των Φίλων σήμερα μαζί μας και βεβαίως ε, την μέλη της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και τα μέλη της Μικτής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ενώσης Τουρκίας είναι παρόντα. Χαίρομαι που είναι κοινή αυτή η πρωτοβουλία και χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε εδώ κυρία μου. Όσον αφορά τη δική μας Επιτροπή, την Επιτροπή Ισότητας των Φίλων, παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις στην Τουρκία, οτιδήποτε σχετίζεται με τα δικαιώματα των γυναικών, με την ισότητα των φίλων και είναι υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για μας ε, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην Τουρκία. Θα έπρεπε να σας πω ίσως ότι η Επιτροπή μας έστειλε μια αντιπροσωπεία στην Τουρκία το Φεβρουάριο, φέτος, το Φεβρουάριο του 2012 και υιοθετήσαμε και μια έκθεση προοπτική για το 2020 για τις γυναίκες στην Τουρκία. Αυτός είναι ο τίτλος της εκθέσεως. Σημειώνουμε ότι υπήρξαν κάποιες εξελίξεις στην Τουρκία όσον αφορά την πολιτική για την ισότητα των φύλων. Παρ' όλα αυτά ε, θα έλεγα ότι η νομοθεσία δεν εφαρμόστηκε με ισότιμο τρόπο παντού και δεν είμαι σίγουρος ότι ε, η νομοθεσία έχει εφαρμοστεί σε όλα τα μέρη της χώρας ε, και παραμένουν, απομένουν πολλά πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα τομέα. Η ισότητα βεβαίω είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναπόσπαστο τμήμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαι σίγουρο ότι τα μέλη θα σα θέσουν διάφορε ερωτήσει, τα μέλη τη Επιτροπή Ισότητα των φίλων. Αλλά δράτω με τη ευκαιρία τώρα για να σα θέσω αμέσω ε, τρία ερωτήματα, κυρία Ζάνα, αν επιτρέπετε. Υπαριθμόν ένα. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά το γεγονός ότι ελάχιστες γυναίκες συμμετέχουν στην πολιτική στην Τουρκία. Ένα χαμηλό επίπεδο συμμετοχής γυναικών στην πολιτική ζωή. Πιστεύετε επίσης ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του κουρδικού και του ε, τουρκικού πληθυσμού όσον αφορά αυτό το θέμα. Δεύτερον, η βία βάση του φύλου και η βία ε, ανδρών κατά γυναικών, αυτό είναι ένα πρόβλημα και για την Τουρκία και για την Ευρώπη στο σύνολό της. Υπάρχει μια νέα νομοθεσία η οποία υιοθετήθηκε πρόσφατα ε, νομοθεσία, νόμος για να προστατεύσει τις οικογένειες και να αποφευθεί η βία ε, λόγω ε, διαφοράς των ανδρών κατά γυναικών. Ποια είναι η άποψή σα, θα πετύχει καλό αποτέλεσμα αυτό, πιστεύετε ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας θα είναι εύκολη. Και τρίτον και τελευταίο ερώτημα, θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε όσον αφορά τις συζητήσεις που διεξάγονται τώρα στην Τουρκία σχετικά με το δικαίωμα της άμβλωσης και αναφέρομαι στα δικαιώματα τα κοινωνικά και τα αναπαραγωγικά. Λοιπόν, τη συζήτηση για την άμβλωση. Αυτά είναι, αυτοί είναι τρει θεματικοί τομεί που αν είχα την καλοσύνη θα ήθελα να μου απαντήσετε. Προσβλέπω στη συζήτηση και σε περαιτέρω ερωτήσει που σου υποβληθούν από άλλα μέλη. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκούσταυσον. Και τώρα η κυρία Κοπά τη αντιπροσωπεία ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Τουρκία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Λοχμπίλερ. Η συζήτησή μα σήμερα αφορά την ελευθερία του λόγου και τα δικαιώματα των γυναικών στην Τουρκία και στην μεικτή αυτή κοινοβουλευτική επιτροπή είχαμε τη δυνατότητα στις 14 Ιουνίου να συζητήσουμε το θέμα με τον νέο Τούρκο Υπουργό για θέματα γυναικών. πιστεύω ότι είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα για αυτή την επιτροπή διότι έχουμε εδώ σαν βασικό, βασική ομιλήτρια ε, την κυρία Λέλα Ζάνα, βραβείο Ζαχάροφ, που είναι ένα σύμβολο συνεχής πάλης για τα δικαιώματα της γυναίκας, για την ελευθερία της έκφρασης και του λόγου που φυλακίστηκε και υπέφερε πολυπή κύλα εν ονόματι του ε, κουρδικού λαού. Η Λέλα Ζάνα παρουσίασε πρόσφατα ένα σχέδιο σχετικά με τον κουρδικό λαό για να προτείνει πρόθεση της διαθετήσεως του θέματος και συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Ταχύπ Ερντογάν, αυτό θεωρείται πρόοδος και ήταν έτοιμη να δεχτεί ότι ήταν η δημοσία ότι ήταν η μόνη που θα μπορούσε να κάνει βήματα, βήματα για την επίλυση των συγκρούσεων. Ότι ο κ. Ερντογάν θα μπορούσε να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων. Ε, και πιστεύουμε ότι αυτό δείχνει μια κυριότητα και θα μπορούσαμε όλοι να μάθουμε αυτό το παράδειγμα. Λοιπόν, ζητήθηκε μια ειρηνική διευθέτηση και αισθάνονται επικρία οι Κούρδοι ε, και δεν είναι εύκολο να ζητήσει η Λέιλα Ζάνα αυτό το συμβιβασμό, αυτόν τον τρόπο. Η κυρία Λέιλα Ζανά είναι μια καθάρια φωνή με ηθική αικαιρεότητα ε, και τη σέβονται στην κοινότητά της. Είναι η ηθική αικαιρεότητα που ξεπερνά το όλο ιστορικό και την παράδοση και την απονομή βραβείων προς αυτήν. Είναι θετική δύναμη μια γυναίκα που πρέπει να την υπολογίσει κανείς, που αξίζει να επενδύσει κανείς με πολιτική και ηθική υποστήριξη. Διότι κάθε φορά που υποστηρίζουμε ανθρώπους σαν τη Λελά Ζάνα, επενδύουμε στην ειρήνη. Σε λαού που θέλουν να προχωρήσουν στα μισά, του δρόμου παρά τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες. Η Λελά Ζάνα μπορεί να μιλήσει εν ονόματι της ελευθερίας του λόγου, των δικαιωμάτων των γυναικών, εκ μέρου του λαού τη και είναι πρόθυμη να μιλήσει για την ειρήνη. Γι' αυτό θα πρέπει να την ακούσουμε προσεκτικότατα σήμερα. Γι' αυτό η δημοκρατία της Τουρκίας θα πρέπει και εκείνη να την ακούσει. Διότι αν ο κουρδικός λαός χάσει την εμπιστοσύνη του ε, στη Λαϊλά Ζάνα και στις μάχες του Δίνη, δεν θα χάσουν την εμπιστοσύνη του σε ένα πρόσωπο και μόνο σε ένα άτομο, θα χάσουν την εμπιστοσύνη στη διπλωματία και στην πολιτική προσπάθεια. Και η κυρία Ζάνα δεν είναι μόνο σημαντική σαν άνθρωπο, σαν άτομο, αλλά και σαν σύμβολο. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κουρδική κοινότητα δεν είναι απλώς μια μειονότητα που ε, βρίσκεται σε συγκεκριμένη περιοχή και επικρατεί της Τουρκίας. Περισσότεροι ε, Κούρδοι ζουν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη από ό,τι στον Διαμπακύρ. Και ο κουρδικός λαός ε, αποτελεί, έχει διαφορετικές πολλές κοινωνικέ και πολιτικές. Είναι φτωχοί, πλούσιοι, επαγγελματίε, ε, χωρικοί. Ο κουρδικός λαός ε, ζουν σε μια περί... ζει σε περίπλοκη πραγματικότητα και υπάρχει ανοιχτή αντιπαράθεση και είναι αντιπαράθεση του α έναντι του β. Η ειρήνη είναι πιο περίπλοκη από τον πόλεμο και γι' αυτό εκείνοι που δέχονται τον περίπλοκο χαρακτήρα αυτών και είναι έτοιμοι για να βρούνε μια περίπλοκη ρύθμιση εντό δημοκρατικού κράτου με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αξίζουν το σεβασμό μα ή τολμώ να πω ακόμα και το θαυμασμό μα. Δεν είναι εύκολο το μονοπάτι, δεν είναι και το πιο ένδοξο μονοπάτι, αλλά είναι ένα μονοπάτι που έχει διαλέξει η κυρία Λαζάνα για τον εαυτό τη. Και εδώ θα ήθελα να την ευχαριστήσω εκ νέου που είναι εδώ μαζί μας. Thank you, Madam Ευχαριστώ κυρία Κόπα. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Λεϊλά Ζανά και θα ήθελα και εγώ θερμά να σας καλωσορίσω και πάλι. Για μένα προσωπικά ήταν πολύ σημαντικό να σας δω εδώ. Εγώ όταν ήμουν φοιτήτρια έκανα μια εκστρατεία για την απελευθέρωση της Λέιλα Ζανά. Δέκα χρόνια που ήσασταν στη φυλακή όλοι είχαμε ε, <clears throat> ε δείξει τη διαθεσιμότητά μας να πάμε να επισκεφθούμε την φυλακή όπου ήσασταν φυσικά δεν μας άφησαν. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ακούσουμε αυτά τα λόγια σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά όλους για την υποδοχή σας εδώ. Απευθύνομαι προς την Υποεπιτροπή λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ε, προς, την, ε, προς τα μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων της Γυναίκας και Ισότητας των Ευκαιριών, προς τα μέλη της Επιτροπής, της μικρής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Καλημέρα σας. Σήμερα συζητούμε θέματα παραβιάσεων των δικαιωμάτων. Το, στην Τουρκία, στο Κουρδιστάν ε, αντιμετωπίζουν άνθρωποι πολύ σημαντικές ε, διώξεις, πιέσεις, γυναίκες και παιδιά βρίσκονται κρατούμενοι στις φυλακές, ε, στερούνται βασικά δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αναπαλωτρία τα δικαίωματα που απορρέουν από τη φύση και μόνο του ανθρώπου και απαιτούν αξιοπρεπή διαβίωση, συνιστούν ένα δικαίωμα σε αξιοπρεπή διαβίωση και αντιμετώπιση ωστόσο και δεν μπορούν να υπαχθούν σε οποιαδήποτε ε, ιδέα ή ε, όφελος δημόσιο, οικονομικές αξίες ή πολιτικές αξιολογήσεις. Είναι η δυνατότητα για τον άνθρωπο να ζει όπως το εννοεί ο ίδιος, να διαμορφώνει μόνος τη ζωή του. Σήμερα, οι συνθήκες διαβίωσης στις οποίες βρισκόμαστε, μέσα από ε, κρυφούς πολέμους, από αυταρχικά πολιτεύματα, από κατασταλτικά καθεστώτα, δίνουν μια εικόνα ενός σκληρού δρόμου, ενός μακρύ δρόμου και υψηλών τυχών που πρέπει να περάσει κανείς για να βρεθεί στην διεκδίκηση των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Εμεί προσπαθούμε πάντοτε να κάνουμε να ακούγεται η φωνή μας και το στόχο αυτόν τον υλοποιούμε απευθύνοντας το λόγο και σε εσάς και αυτό θέλω να σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε. Δυστυχώ όμως πρέπει να πω ότι στην Τουρκία, στο Κουρδιστάν, οι παραβιάσεις των ανθρωπινών δικαιωμάτων είναι παρούσες, τις διαπιστώνουμε καθημερινά και ανεξαρτήτως της ε, προέλευσης της ε, κοινωνικής τάξης, της φυλής, ε, βλέπουμε να γίνονται παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είτε πρόκειται για δημοσιογράφους, για συγγραφείς, ε, για εκδότες, πανεπιστημιακούς, φοιτητές, συμμαθητές, ε, καλλιτέχνες, για συνδικαλιστές, πολιτικούς, συμβουλευτέ ή για τοπικούς ερετούς άρχοντες. Βλέπουμε ότι διώκονται, συλλαμβάνονται, δικάζονται και καταδικάζονται από τα δικαστήρια για μεγάλο χρονικό διάστημα και συστηματικά με εντολές της ε, αστυνομίας συλλαμβάνονται και βρίσκονται κρατούμενοι και ανακρίνονται ε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην Τουρκία και δυστυχώς ε, αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα παραβιάσεως των ανθρωπινών τους δικαιωμάτων. Αυτό συνέβη. Συνέβαινε και στο παρελθόν, συνέβη και τώρα. Το μήνα που περάσαμε μόλις ξεκίνησε μια στάση κρατουμένων στην Ούρφα, σε μια φυλακή τύπου ε, όπως ονομάζεται, από 13 κρατούμενους, οι οποίοι ε, από τους κρατούμενους ύστερα από με αποτέλεσμα το θάνατο 13 κρατουμένων και που στη συνέχεια επεκτάθηκε στις φυλακές του Άντεπ, των Αδάνων, του Καραμάν. Ήταν μια στάση ε, αντίδρασης ε, στις συνθήκες διαβίωσης στη φυλακή της Σούρφα. Ήταν άνθρωποι που καταδικάστηκαν το 2010 και το 2011 ε, δεν άντεξαν τις συνθήκες διαβίωσης και έβαλαν φωτιά στα κελιά τους. Έχουμε να κάνουμε με φυλακές όπου 300 άτομα συμβιώνουν, ε, σε χώρο μάλλον 300 ατόμων συμβιώνουν πάνω από 1000 άτομα. Έχουμε να κάνουμε με τριπλάσιο αριθμό κρατουμένων και βέβαια ε, υπέρβαση κάθε ορίου ανθρώπινης διαβίωσης. έχει διαπιστωθεί και από το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, και από τη Διεθνή Αμνηστία ότι οι συνθήκες κράτησης και διαβίωσης στις τουρκικές φυλακές είναι πολύ κακές, είναι υπερβολικά μεγάλος ο αριθμός και η συγκέντρωση κρατουμένων μέσα σε μικρούς χώρους και οι συνθήκες κράτησης δεν αντιστοιχούν στα ανθρώπινα, δικαιώματα και οδηγούν σε προβλήματα, σε στάσεις ακόμη και σε φόνους. Αντί για 80.000 κρατουμένους στις φυλακές Τουρκίας ε, αυτή τη στιγμή βρισκόνται 130.000 και άνω κρατούμενοι. 120.000 από αυτούς είναι κρατούμενοι για λόγους ποινικούς, 9.000 για λόγους πολιτικούς και πάνω από 2.000 από αυτούς κρατημένους είναι για οργανωμένο έγκλημα, μαφία κτλ. Το προσωπικό στις φυλακές είναι ανεπαρκές και βέβαια προξενεί ανησυχίες η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται. Τα δικαιώματα των κρατουμένων παραβιάζονται και ως προς τις συνθήκες της ε, υγιεινής, της επικοινωνίας ε, ή της ασφάλειάς τους. Είναι πολλές οι περιπτώσεις των ε, βιοπραγιών και των βιασμών ακόμη 2.500 παιδιά πρέπει να σας πω και νέοι βρίσκονται στις φυλακές μας και κινδυνεύουν από αυτές τις βιοπραγίες και τους βιασμούς. 5.000 περίπου γυναίκες ε, δεν είναι σε θέση να διατυπώσουν ούτε καν μία προσφυγή ή διαμαρτυρία για τις συνθήκες κράτησής τους. Παιδιά δε σε ηλικία 0 έως 6 ετών είναι άνω των 300 στις τουρκικές φυλακές γιατί μένουν ε, μαζί με τις μητέρες τους. Αλλά δεν έχουν τις, ε, τη δυνατότητα της πρόσβασης υπηρεσίας που θα έπρεπε να έχει ένα παιδί στην κατάσταση αυτή. Τα δε προβλήματα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οι γυναίκες στις ε, συνθήκες κράτησης στην Τουρκία επηρεάζουν πολύ συχνά ακόμα και την υγεία τους ε, με συνέπειες, ε, σε συνέπειες σοβαρές ασθένειες γυναικολογικού τύπου όπως ε, καρκίνο του, της μήτρας, του στήθους και ούτω καθεξής, του μαστού και το καθεξής. Ταυτόχρονα δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι οι γυναίκες κρατούμενες υφίστανται γυναικολογικές εξετάσεις σε περίπτωση αρρώστιας από τους άντρες δεσμοφύλακες στις φυλακές. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με ένα παρελθόν, με μια κληρονομιά βαριά που έχει αφήσει η Χούντα της 12 η Σεπτεμβρίου. Και ξεκολουθούν στις φυλακές του Διάρμπακερ, του Μάμακ, του Μέτρης να ε, πραγματοποιούνται, να διαπράττονται τα εγκλήματα που έχουμε δει ε, τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν έχουν σταματήσει. Παραδείγματι βλέπουμε ότι το 1996 σφαγιάστηκαν δέκα κρατούμενοι και μέχρι σήμερα δεν έχει αποκαλυφθεί ποιος ήταν υπέτειος, δεν έχει κανείς προσαχθεί στην δικαιοσύνη. Θα ήθελα να μου επιτρέπετε τώρα να σας κάποια στοιχεία για τις συνθήκες κράτησης των γυναικών στην Ούρφα. Τα παιδιά, καταρχάς, τα παιδιά τα οποία είναι γνωστά στην κοινή γνώμη της Τουρκίας ως τα παιδιά που λιθοβολούν, τα παιδιά που πετάνε πέτρες, ε, που διαμαρτυρήθηκαν δηλαδή στους δρόμους, είναι παιδιά 12 με 18 ετών περίπου και ε, βρίσκονται εκτεθειμένα στις φυλακές σε κάθε τύπου βίας ε, και βιοπραγία και εκμετάλλευση. Στο ε, κρατητήριο στη φυλακή του Ποζάντη έχουν, ε, για το κρατήριο μάλλον του Ποζάντη έχουν ακουστεί πάρα πολύ ε, δυσάρεστες και ανησυχητικέ πληροφορίες για τέτοιου είδους βιοπραγίες, ακόμη και βιασμούς. Βλέπουμε ότι το κράτος δεν είναι διατεθειμένο να κυρώσει να διώξει και να κυρώσει αυτές τις ε, πράξεις, αυτά τα δικήματα εις βάρος των κρατουμένων και αυτό ισοδυναμεί με επικύρωση τους, με έγκριση τους. Έγιναν ε, στην ε, φυλακή του Ποζάντ επεμβάσεις από τις, φυλακές, από τις αστυνομικές αρχές οι οποίες ακόμη περισσότερο επιδίνωσαν τις συνθήκες αντί να εξασφαλίσουν προστασία των κρατουμένων παιδιών. Πρέπει να αναπτυχθεί λοιπόν ένα σύστημα διαφανές ελέγχου των συνθήκων κράτης των φυλακών. Πρέπει να υλοποιηθεί ουσιαστικά το πρωτόκολλο για την απαγόρευση των βασανιστήριων και να θεσπιστεί ο προβλεπόμενος μηχανισμός και πρέπει η Γενική Αμνηστία που είχε από το 1974 να δοθεί επιτέλους να ανακηρυχθεί. Πρέπει να πω ότι στη ζωφερή αυτή η εικόνα που παρουσιάζουν τα κρατητήρια, τα σοφροναστικά είναι στην Τουρκία, τη συμπληρώνουν κακές, εσφαλμένες και ε, προβληματικές, ελαττωματικές αποφάσεις των δικαστηρίων. Πρέπει να πω ότι εμείς έχουμε πολλά πράγματα να πούμε μόνο και μόνο ε, για τις προσβολές, ε, τις απειλές, ακόμα και τις επιθέσεις που έχουμε υποστεί όταν χρησιμοποιούμε την γλώσσα μας, την κουρδική γλώσσα. Έχουμε μάθει να ζούμε με αυτή τη βία και αυτές τις απειλές, αλλά πρέπει αυτό πια να σταματήσει, πρέπει αυτή η βία να απαγορευτεί και να αναγνωριστεί ως κάτι το κακό. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αποδεκτή αυτή η κατάσταση από το τουρκικό κράτος. Και άλλο ένα παράδειγμα που έχω να σας δώσω είναι αυτό της δίκης της ε, περίφημης ε, Νετσέ με ενός κοριτσιού 13 ετών που έπεσε θύμα πολλαπλών ε, και επαναλαμβανόμενων βιασμών από ομάδα αντρών στους οποίους συγκαταλέγονταν και δημόσιοι λειτουργοί και για τους οποίους εκρίθη ότι η κοπέλα ήταν σε συνένεση και πλήρη επίγνωση της καταστάσεως και ως εκ τούτου αναγνωρίζονται ελαφρυντικά στοιχεία στην υπόθεσή της. Έτσι τιμωρήθηκαν με χαμηλότερες ποινές. με τις νέες προτάσεις για την αναθεώρηση της δικαιοσύνης ε, και την αλλαγή του καθεστώτος των ε, δικαστηρίων ειδικών εξουσιών όπως ονομάζονται δεν αλλάζει το πρόβλημα, ε, δεν αντιμετωπίζεται, είναι μόνο παρηγορητικής λειτουργίας αυτά τα μέτρα. Χρειάζεται ριζική αλλαγή του μηχανισμού της λειτουργίας της δικαιοσύνης στην Τουρκία. Οι δε οικουμενικές αξίες των δικαιωμάτων είναι ε, συμπεριλαμβάνουν και το αυτονόητο για άλλους ε, στον κόσμο δικαίωμα της επιλογής, της εκλογής του ηγέτης Του ηγέτης τους. Είναι για τον Κούρδο μεγάλο πόνο το γεγονό ότι ο ηγέτης τους, ο, Τζαλάς, ο Τζαλάν, βρίσκεται στη φυλακή και στην απομόνωση. Ζητούμε από αυτό λοιπόν να κάνει ε, στο θέμα αυτό ό,τι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και σημειώνουμε ότι ο, ο Τσαλάν ήδη είχε προσπαθήσει ε, διαφεύγοντας από την Τουρκία και στο παρελθόν να δώσει ευκαιρίες για διάλογο, είχε δηλώσει ότι ήταν έτοιμος για διάλογο. Η Ευρώπη όμως δεν μπόρεσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και της εποχής και έτσι Τώρα, με τις συνθήκες που αντιμετωπίζουμε και την κράτηση στην απομόνωση του Τσαλάν, περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον να αναλάβει τις ευθύνες της και να δραστηριοποιηθεί στην υπόθεση αυτή. Πρέπει να επαναλάβω ότι η κοινωνία είναι έτοιμη πια για λύσεις. Πρέπει μόνο η πολιτική εξουσία να λάβει το θάρρος και να πράξει τα απαραίτητα. Στις συνθήκες ε, τη προστασία ή τη λειτουργία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στην κοινωνία, ακόμη δυστυχώ έχουμε πολλά προβλήματα. Ε, παραμένουν προβλήματα ω προ την ισότητα ανδρών και γυναικών. Ε, είναι ακόμη περιορισμένη η εκπροσώπηση των γυναικών ε, και παρά τις πολλές προσπάθειες και τους αγώνες που έχουν γίνει δεν έχουμε μπορέσει να ανατρέψουμε το δυσάρεστο πίνακα που παρουσιάζεται από τις ειδήσει που παίρνουμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωση, μόνο τον Ιούνιο, τον μήνα που μόλις μας πέρασε, είχαμε 7 φόνους εις βάρος ε, γυναικών και παιδιών, 9 σωματικές ε, βλάβες εις βάρος γυναικών, 8 βιασμούς εις βάρος γυναικών, 12 ε, σεξουαλικές παρενοχλήσεις εις βάρος γυναικών και πολλά θύματα, τα περισσότερα από τα θύματα έπεσαν θύματα στα χέρια των ε, συζύγων τους ή ανδρών της, ε, του κύκλου τους, του, στενού οικογενειακού του ε, κύκλου. Για το 2012 τα στοιχεία είναι ότι δολοφονήθηκαν 78 γυναίκες, 116 γυναίκες έπεσαν θύματα βία, 49 γυναίκες θύματα βιασμού, 88 γυναίκες σεξουαλικής παρενόχλησης. Το πιο επώδυνο από τα στοιχεία όμως είναι ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης ε, σημειώνει στις στατιστικές του ότι από το 2002 στο 2009 η αύξηση των εγκλημάτων εις βάρος των γυναικών ήταν της τάξης του 1400%. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολη η κατάσταση, ιδιαίτερα δε για τις γυναίκες ε, ε, που έχουν πολύ χαμηλή δυνατότητα συμμετοχή στην αγορά εργασίας, την ε, παιδεία, να απασχόληση γενικότερα και την ε, κοινωνική ε, και χαμηλή δυνατότητα πρόσβαση στην κοινωνική πρόνοια. Είμαστε υποχρεωμένοι γι' αυτό για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στην παιδεία, στην απασχόληση, στην κοινωνική πρόνοια, να μιλάμε τουρκικά και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για μας. Χρειαζόμαστε, χρειάζονται πολλές φορές οι γυναίκες οι οποίες μόνο τη μητρική τους γλώσσα γνωρίζουν να χρησιμοποιήσουν ως διερμηνέα έναν ε, άντρα του κύκλου τους ε, για να λύσουν κάποιο πρόβλημα που έχουν. Πράγμα το οποίο βέβαια επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τον έλεγχο μπορεί να ασκήσει ένας άντρας σε μια γυναίκα. Σε πολλές περιπτώσεις ε, χρησιμοποιούνται δύο γλώσσες διαφορετικές ε, μέσα στο ίδιο σπίτι, γιατί οι γυναίκες μπορεί να καταλαβαίνουν με τα τουρκικά αλλά δεν μπορούν να τα μιλήσουν, ε, τα παιδιά να καταλαβαίνουν με τα κουρδικά αλλά μην μπορούν να τα μιλήσουν και έτσι επιδεινώνεται το χάσμα μεταξύ των γενναιών και σε γλωσσικού όρου. Υπάρχει, ένα, υπάρχει όμως ε, μια θετική εικόνα σε όλα αυτά, ότι οι γυναίκες στον αγώνα τον κουρδικό, στον, στην, στο κουρδικό κίνημα έχουν λάβει το ρόλο που τους αξίζει, έχουν διεκδικήσει ε, ουσιαστικά δικαιώματα και τα έχουν επιτύχει, έχουν διεκδικήσει το μέλλον τους δηλαδή. Πρέπει να ακούσουμε τα αιτήματα που διατυπώνονται από όλες αυτές τις ε, οργανώσεις των γυναικών που αγωνίζονται για το κουρδικό θέμα και να τις στηρίξουμε. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία νομίζω θα ήταν να ε, θεσπιστεί Υπουργείο για θέματα των γυναικών. Αυτό είναι απαραίτητο. Και περιμένουμε επίσης ε, να ε, αναφερθώ τώρα σε μια πληγή εμάσουσα ακόμα στο Κουρδιστάν, την πληγή των ανεξιχνίαστων ακόμη φόνων. Είναι από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε τα στοιχεία, ε, περίπου 3.000 οι τα άγνωστα θύματα αυτών των των φόνων που βρίσκονται θαμμένα σε μαζικούς στάφους στις ε, περιοχές μας. 17.500 συνολικά είναι τα ε, θύματα αυτών των των εγκλημάτων. Και θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στην περίπτωση της σφαγής του Ρομπόσκι. Πριν από έξι μήνες ε, ένα αεροπλάνο του τουρκικού στρατού, ένα F-16, ε, άνοιξε πυρά και σφαγέ σε 34 ε, νέους Κούρδους. Προσπάθησε η κυβέρνηση, προσπάθησαν με την παρέμβασή τους αμέσως να συγκαλύψουν το περιστατικό και να μην αποκαλυφθούν τα στοιχεία, αλλά το πρόβλημα υπάρχει, η σφαγή έλαβε χώρα και πρέπει να διερευνηθεί. Έχουν χάσει τη ζωή τους άνθρωποι, έχουν οικογένειες και πρέπει να φτάσουμε πια στο επίπεδο της αποκάλυψης αλήθειας, της διαφάνειας για να μπορέσουμε και να θεραπεύσουμε τις πληγές μας. Παρακαλώ λοιπόν για το θέμα αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλυφθεί ρόλος ενεργός για να διαρευνηθεί η υπόθεση και να αποδοθεί δικαιοσύνη όπως πρέπει. Εν τέλει, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο τελευταίο και σοβαρό ζήτημα. Η ιστορία μας έχει αποδείξει ότι κανένας πόλεμος δεν συνεχίζει ε, επαόριστον. Πρέπει κάποια στιγμή να δοθεί η δυνατότητα για λύση, για συνενώσει και συμφιλίωση μεταξύ των εμπολέμων πλευρών. Αλλά δυστυχώ εμεί στην Τουρκία δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να βρούμε τον τρόπο και τι εσωτερικέ δυναμικέ για να καταλήξουμε σε αυτή τη λύση. Σε αυτό θα ήθελα να στήσω πάλι τη βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί πιστεύουμε ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει οικονομικά κέρδη και συμφέροντα, αλλά περισσότερο από αυτά η Τουρκία χρειάζεται δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερίε και εν τέλει χρειάζεται βιώσιμη ειρήνη. Και γι' αυτό παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει λάβει πρωτοβουλίες και δραστηριότητα έτσι ώστε να δούμε μια πραγματικότητα, ώστε να δούμε μια ζωντανή λύση. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ και πάλι το Πρόεδρο. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ, Λαϊλά Ζανά, για την πάρα πολύ λεπτομεριακή σας παρουσίαση για την κατάσταση των σοφρονιστικών καταστημάτων στην Τουρκία. Τονίσατε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να εφαρμοστούν και στην πράξη και θα πρέπει να δούμε τι είδους θεσμοί υπάρχουν στην Τουρκία που μπορούν να αναλάβουν αυτό το έργο. Και όπως είπατε στο τέλος, θα πρέπει να λάβουν χώρα οι απαραίτητες έρευνες <clears throat> για τους σωματικούς τάφους που έρχονται στο φως τώρα. Αυτό είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο και μια ουσιαστική συμβολή στην διαδικασία ειρήνευσης και συμφιλίωσης για τις οικογένειες ιδίως των θυμάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της συμφιλίωσης που πρέπει να λάβει η χώρα. Δίνω το λόγο τώρα στους βουλευτές γιατί έχουμε χρόνο για να συζητήσουμε. Ίσως μπορούμε να ακολουθήσουμε την εξή ε, διαδικασία. Μαζεύουμε ένα αριθμό από και απαντάτε ομού σε όλους τους ερωτώντες. Έχω τον κύριο Χατζηγεωργίου καταρχήν στον κατάλογο μου. Καλημέρα σας. Καλωσορίζω και εγώ την κυρία Ζανά στο Κοινοβούλιο. Θα μου επιτρέψετε καταρχήν να εκφράσω τη λύπη μου γιατί ενώ εδώ βρίσκομαι ως μέλος της Μιχτής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, όπου πολλά μέλη αυτής της Επιτροπής εκφράζουν συχνά πυκνά την εντύπωση ότι η δημοκρατία στην Τουρκία ανθίζει μέρα με τη μέρα. Ε, στην παρούσα συνεδρία δεν βλέπω παρά μόνο ίσως δύο-τρία μέλη αυτής της Επιτροπής. Γι' αυτό θα παρακαλούσα, εάν είναι δυνατόν, η ομιλία σας να σταλεί στα email μάλλον όλων των Ευρωβουλευτών του Κοινοβουλίου. Ε, έχω μία εντύπωση και μία ερώτηση. Πιστεύω ότι ε, χιλιάδες προβλήματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί το γεγονός ότι το ΠΚΚ έχει ονομαστεί τρομοκρατική οργάνωση ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη. Η ερώτησή μου είναι αν πράγματι, αν και εσείς ε, έχετε την ίδια εντύπωση ότι χιλιάδες δηλαδή παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν να κάνουν με την χρησιμοποίηση του γεγονότος ότι το ΠΚΚ χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση και έχω και μια δεύτερη ερώτηση. Θέλω πάρα πολύ καθαρά και ίσα να σας ρωτήσω εάν εσείς θεωρείτε ε, αυτή την οργάνωση τρομοκρατική και γιατί. Thank you. Uh, and just... Ευχαριστώ. Από τη δική μου οπτική γωνία βλέπετε πόσοι βουλευτές είναι παρόντες. Είναι 12 βουλευτές από ό,τι βλέπω, αλλά δεν τους βλέπω όλους γιατί πολλοί είναι εκτός του οπτικού μου πεδίου. Για την παρουσίαση τώρα της ε, Λεϊλά Σανά, που είναι και βραβείο Σαχάροφ, εμείς έχουμε και άλλες συναντήσεις μέσα στην ημέρα σήμερα με τη δική αυτή ομάδα για την υποστήριξη του βραβείου Σαχάροφ. Νομίζω θα ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα να υπάρξει διανομή, όπως είπατε, της παρουσίασης της κυρίας Λεϊλά Σανά σε όλους τους βουλευτές. κυρία Μπάουερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ θέλω να χαιρετήσω την παρουσία της κυρίας Λέιλα Σανά και όταν ξέραμε εμεί ότι πάλι έχετε καταδικαστεί από τα τουρκικά δικαστήρια κάναμε πολλές διαμαρτυρίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δύο ερωτήματα. Είπατε ότι υπάρχουν και πάλι προβλήματα με, το, με τη χρήση της κουρδικής στο σχολικό σύστημα και την χρήση στα σχολεία. Πριν από λίγα χρόνια άνοιξαν σχολεία στα κουρδικά, αλλά είπατε ότι τα παιδιά δεν πηγαίνουν σε αυτά τα σχολεία. Επίσης, ε, γενικά αν υπάρχουν προβλήματα με τη χρήση της κουρδικής θα ήθελα να ξέρω από τη δική σας πλευρά. Ένα δεύτερο θέμα είναι η λεγόμενη φόνη τιμής. Είπατε ότι η βία κατά των γυναικών αυξάνεται ο αριθμός των βιαίων πράξεων κατά των γυναικών αυξάνεται συνέχεια. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η κατάσταση με τους φόνους για λόγους τιμής. Όταν ήμασταν στην Τουρκία, ακούσαμε ένα εμπειρογνώμονα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο οποίος μας είπε ότι μειώνεται ο αριθμός των φόνων τιμής στην Τουρκία. Με αυτά όμως που είπατε εσείς, έχω την εντύπωση ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο για τους φόνους τιμής. Η κυρία Κιλ Νίλσεν. Σας ευχαριστώ. Το ερώτημά μου θα είναι πολύ σύντομο, κυρία Ζανά. Συναντήσατε πρόσφατα τον Πρωθυπουργό Ερντοάν. Θα μπορούσατε να μας πληροφορήσετε ίσως για τις θετικές προοπτικές οι οποίες προέκυψαν από αυτή τη συνάντηση. Σας ευχαριστώ. Έχω άλλους οκτώ συναδέλφους, αλλά θα δώσω τώρα το λόγο στη Λέιλα Σάνα για να απαντήσει την πρώτη σειρά ερωτήσεων. Το μεγαλύτερο, το πιο επώδυνο πρόβλημα είναι αυτό της ε, γλώσσας. Αυτό είναι που με απασχολεί πιο πολύ εμένα και με αυτό θα ξεκινήσω. Δεν υπάρχει μέρος στον κόσμο όπου ένας λαός να έχει υποστεί αυτή την απαγόρευση της χρήσης της γλώσσας του. Πριν από 32 χρόνια, στις 12 Σεπτεμβρίου, με, την, με το στρατιωτικό πραξικόπημα, εισήχθη ένα σύστημα καταπίεσης εις βάρος ενός λαού, άρνησης ταυτότητάς του, απαγόρευσης της γλώσσας τους αν διανοηθείτε ότι έχουν περάσει 32 χρόνια και από τότε θα αντιληφθείτε. Θυμάμαι πολύ καλά. 7 η ώρα το πρωί πηγαίναμε στις πόρτες των φυλακών. Περιμέναμε μέχρι το βράδυ, μέχρι τη νύχτα, για να δούμε τον άνθρωπό μας για ένα λεπτό. Ένα λεπτό ακριβώς. Και μέσα σε αυτό το ένα λεπτό, στην ε, καμπίνη επικοινωνίας που έχουμε στις φυλακές, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε κουρδικά. Εγώ δεν μπορούσα τότε τη σκέψη μου να τις εκφράσω στα τουρκικά. Καταλάβαινα, αλλά δεν μπορούσα να εκφραστώ όπως ήθελα. Τώρα φανταστείτε ότι μέσα από αυτές τι επισκέψει φυλακέ έμαθα εγώ τουρκικά. Εξαιτία αυτών των επισκέψεων. Άρνηση λοιπόν και απαγόρευση τη γλώσσα ενό λαού. Και σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει άλλο μέρος στον κόσμο όπου μπορεί να στείλουμε τα παιδιά μα στο σχολείο και να μην έχουμε αρκετά λεφτά για να τους βάλουμε στην τσέπη ε, το κολατσιό τους, τα λεφτά αυτά τα οποία θα, πρέπει, θα πρέπει να έχουν πάει στην εκμάθηση της γλώσσας. Γιατί μας είπαν ότι δεν έχουν λεφτά η κυβέρνηση να κάνει μαθήματα κουρδικής και τα κλείσανε τα, τα τμήματα. Ή όπου υπάρχουν τα έχουν κάνει μάθημα επιλογής σε μια ξένη γλώσσα. Διότι εμείς δεν είμαστε ένας λαός ο οποίος να ζει με δικαιώματα ενός λαού που ε, έχει εγκατασταθεί και ζει σε μια περιοχή. Ιστορικά δεν είναι γνωστό πότε εμφανίστηκαν οι Κούρδοι στην περιοχή μας. Είναι πολύ αρχαίος λαός, αλλά από την ε, ίδρυση του τουρκικού κράτους και από την ίδρυση του τουρκικού κράτους πάντοτε οι Κούρδοι έχουν συμβάλει σε αυτό το κράτος θετικά, έχουν αγωνιστεί για να το στηρίξουν. Πρέπει λοιπόν η κουρδική γλώσσα να είναι γλώσσα της εκπαίδευσης, της βασικής εκπαίδευσης για να μην χαθεί, για να μπορούμε να τη συζητούμε. Και αυτό που υπενήχθηκα ε, μέσα από τη συζήτηση, από την ομιλία μου, είναι ότι η διάδοση του κουρδικού πληθυσμού είναι τέτοια που οι μισοί Κούρδοι βρίσκονται τώρα στη δυτική Τουρκία, δηλαδή στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια. Αυτοί δεν γνωρίζουν πια την κουρδική γλώσσα. Τα παιδιά του δεν την έχουν μάθει, δεν τη μιλάνε σε μετρική γλώσσα. Και έτσι χάνεται αυτό ο διάλογο χάνεται αυτή η δυνατότητα της επικοινωνίας. Πράγμα το οποίο επιδεινώνει και το χάσμα και την αντιπαράθεση μεταξύ των γενναιών. Η, η μάνα όταν προσπάθησα να εξηγήσω άλλωστε και με την, ομιλία, με την ομιλία μου, εάν πρέπει να μιλήσει σε κάποιο φορέα δημόσια αρχή, είναι υποχρεωμένη να συνοδεύεται από τον άντρα της ή από τα παιδιά της για να τη βοηθήσουν να τις μεταφράσουν. Αυτό επιφέρει ε, ανισότητα στις ευκαιρίες, στις δυνατότητες. Και εάν η αφομοίωση είναι, όπως είχε πει ο Πρωθυπουργό μας, έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, τότε πρέπει αυτό το ζήτημα που το βλέπουμε εμείς καθημερινά να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά και να περάσει στη βασική εκπαίδευση η διδασκαλία της κουρδικής γλώσσας. Σε πολλές περιοχές του Κουρδιστάν αυτή τη στιγμή, μέχρι και στα πιο μικρά χωριά έχουν φτιάξει σχολεία. τα παιδιά μπορούν να μιλάνε τα κουρδικά σαν μητρική γλώσσα μόνο μέχρι τα... μπορούσαν μέχρι τώρα να μιλάνε μέχρι τα 7 τους χρόνια, μέχρι να πάνε δηλαδή στο δημοτικό. Τώρα έχει αρχίσει η υποχρεωτική εκπαίδευση από τα 5 χρόνια από την υπηαγωγείο και άρα ήδη από τα 5 χάνεται η κουρδική ως μητρική γλώσσα. Σε αυτό πρέπει να διδοθεί ιδιαίτερη, να επιδειχθεί ιδιαίτερη ευαισθησία και ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με κάθε ευκαιρία που μας δίνεται. Έχουν γίνει τόσες ε, δηλώσεις, ε, τροποποιήσεις, κανονισμοί, ψηφίσματα για τη μητρική γλώσσα, για το δικαίωμα της μητρικής γλώσσας και όμως αυτό τα προβλήματα τα δικά μας δεν τα έχει λύσει. Και έτσι έχει εισαχθεί η κουρδική σαν μια κατεπιλεγή, κατεπιλογή ε, δεύτερη γλώσσα στα σχολεία. Σε αυτό εγώ δεν έχω αντίρρηση. Όποιος, θέλει, όποιος Τούρκος θέλει να μάθει κουρδικά, πολύ ευχαρίστως, χαρά θα μας κάνει να μαθαίνουν και οι Τούρκοι τα κουρδικά. Αλλά η δική μας μητρική γλώσσα πρέπει να είναι, μια, είναι η γλώσσα της εκπαίδευση, η βασική γλώσσα. Γιατί δεν μπορεί η μία γλώσσα να αντικαταστήσει την άλλη. Δεν υπάρχει περίπτωση να επικαλύψει, να αντικαταστήσει επαρκώ η δευτερεύουσα γλώσσα, την μητρική γλώσσα. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να γίνουν σημαντικά βήματα τώρα. Δεν αρκούν οι μικρέ και παρηγορητικού τύπου λύσεις. Δεν μπορεί μόνο ε, ε, Ούτε καν να, να κλείσουν προσωρινά τις, τις πληγές δεν αρκούν αυτές οι λύσεις πλέον. Πρέπει να δοθούν ουσιαστικές λύσεις και αυτό το λέω όχι μόνο εκ μέρους του έξονόματος του κουρδικού λαού, το λέω εκ μέρους των, του, της Τουρκίας ολόκληρης. Πιστεύω δηλαδή ότι πολλά από τα προβλήματα της Τουρκίας οφείλονται στις παραβιάσεις των ανθρωπινών δικαιωμάτων, των ελευθεριών, της δυνατότητας για πρόοδο και αυτοδιάθεση του ανθρώπου. η βία εις βάρος των γυναικών. Απορρέει πιστεύω περισσότερο από την από την έλλειψη εκπαίδευσης, μόρφωσης. Και Άννα μάθουν οι άνθρωποι να ζουν χωρίς να κάνουν διάκριση μεταξύ πατέρα-μητέρας, μεταξύ κοριτσιού-αγοριού στην οικογένεια. Εάν δηλαδή η εκπαίδευση, η μόρφωση που θα δοθεί στις οικογένειες, στα παιδιά, είναι μόρφωση που έχει εστιάσει στον άνθρωπο και όχι στο φίλο, εάν δοθεί αξία στην ανθρώπινη υπόσταση και όχι στο φίλο, τότε είμαι βεβαία ότι δεν θα έχουμε πια τέτοια φαινόμενα μαζικής βίασης βάρος των γυναικών. και αν όπως συμβαίνει στην κοινωνία η γυναίκα δεν αντιμετωπίζεται ως άνθρωπος, ως ανθρώπινο όνο, τότε προφανώς και θα επιδεινώνονται τα φαινόμενα της βίας της βάρος των γυναικών. Χρειάζεται η μόρφωση λοιπόν. Χρειάζεται η μόρφωση για την πρόοδο και πρέπει να σας πω ότι σε κάποια σημεία έχουμε σημειώσει πρόοδο. Δεν μπορώ να πω ότι όλα είναι ρόδινα, αλλά δεν μπορώ ούτε και να πω ότι τα πάντα πάνε προς το χειρότερο. Αλλά όταν, έχει να όταν πρέπει να δοθεί λύση σε προβλήματα των γυναικών, δεν καταλαβαίνω πώ είναι δυνατόν άντρε, ηγέτε, πολιτικοί να κάθονται γύρω από ένα τραπέζι για να δώσουν λύση στα προβλήματα των γυναικών. Να μην υπάρχει δηλαδή γυναίκα στο τραπέζι αυτών διαπραγματεύσεων. Σε αυτό χρειάζεται να αλλάξουμε νοοτροπίε και στάση. Γιατί ο άντρας που θα κάτσει να συζητήσει αυτά τα ζητήματα δεν θα κοιτάξει τη γυναίκα σαν ε, ισότιμο άνθρωπο, ε, σαν ε, ένα ανθρώπινο που έχει τα ίδια δικαιώματα μαζί του, αλλά μόνο σαν ένα είδου καλοπάτι πάνω στο οποίο θα πατήσει για να ανέβει αυτός πιο πολύ στη ζωή του, για να έχει αυτός περισσότερη πρόοδο και προκοπή. Γι' αυτό νομίζω ότι η Επιτροπή των Γυναικών και το Ισότητα των Ευκαιριών μπορεί, των ευκαιριών μπορεί να συμβάλλει τα μάλα στην υπόθεση αυτή ή πάντως μπορεί να αναλογιστεί δυνατότητες για λύση, γιατί το να λαμβάνονται αποφάσεις για τις γυναίκες, το όνομα των γυναικών, ε, δεν μπορεί να αποτελέσει λύση. Πρέπει η γυναίκα μόνη της να είναι εκείνη η οποία θα διαμορφώσει τις λύσεις και τον τρόπο υλοποίησης ε, των διεκδικήσεών της μέσα των αγώνα της. Γιατί αν ο άντρας δεν μάθει να ε, αναγνωρίζει τη γυναίκα σαν ισότιμο ανθρώπινο, δεν πρόκειται ποτέ να λυθεί το πρόβλημα. Πάντα θα βρίσκεται σε αντιπαράθεση στο γυναικείο με το αντρικό φύλλο και πάντα θα επιδεινώνονται τα προβλήματα ακόμα και της βία στους των γυναικών. Η βία βέβαια είναι πάντα πολύ κακό πράγμα για κάθε κοινωνία, αλλά στην ε, Μέση Ανατολή είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα γιατί εν γέννη οι γυναίκες θεωρούνται ως ένα μηδενικό, δεν υπολογίζονται καθόλου. Μένουν μέσα σε τέσσερις τείχου στο σπίτι ή χαρακτηρίζονται μόνο με την ιδιότητα της μητέρας παίρνουν μια στάμπα δηλαδή μητέρα και εξαντλείται σε αυτό η ύπαρξή τους. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ περιορισμένες δυνατότητες για τις γυναίκες και οι ευκαιρίες μπορούν να τους προσφέρονται. Τα τελευταία 10-15 χρόνια στην Τουρκία βεβαίως πρέπει να πω ότι έχει σημειώσει κάποιες πρόοδες ο αγώνας για την αχειραφέτηση των γυναικών, πρέπει να το πω αυτό. Ναι, βεβαίω το 1934, το 1934 δόθηκε το δικαίωμα τη ψήφου στι γυναίκε. Αλλά αυτό δεν ε, λύνει όλα τα προβλήματα. Τώρα πρέπει να ε, σημειώσουμε ότι ο αγώνα για τη χειραφέτηση των γυναικών έχει επιφέρει κάποιε προόδου, αλλά δεν αρκούν και γι' αυτό ε, έδωσα τα στοιχεία που έδωσα μέσα στην ομιλία μου. Γίνονται, επί παραδείγματι, νομοθετικέ ρυθμίσει, προσαρμογέ στι νομοθεσίε, αλλά δεν αρκούν αυτέ γιατί δεν φέρουν στην ουσία αλλαγή. Για να έρθει στην ουσία αλλαγή ω προ τη θέση των γυναικών, όπω είπα, το μόνο που χρειάζεται είναι μόρφωση εκπαίδευση. αναγκαιο ορο είναι η μόρφωση εκπαίδευση. Μόρφωση εκπαίδευση, αλλά σε κάθε τομέα και στον τομέα ε, στην κατάρτιση επί παραδείγματων των δικαστικών, των αστυνομικών, ε, από το δημοτικό είδε, από το δημοτικό, το παιδί που θα πάει στο δημοτικό σχολείο, αγόρι ή κορίτσι, πρέπει να ε, ακολουθήσει μια, να, να λάβει μια παιδεία που θα αναγνωρίσει την ισότητα των δύο φίλων. Για τις επαφές μου με τον Πρωθυπουργό. Να σας πω, εγώ όπως ήρθα εδώ και σας μίλησα, όπως όταν, είμαι μπροστά όταν μας στα δικαστήρια μιλάω, έτσι μίλησα και στον Πρωθυπουργό. Δεν μπορώ να ε, σας πω πολλές ε, λεπτομέρειες ε, αυτής της συνάντησης τουλάχιστον από πλευρά του Πρωθυπουργού τι υπόθηκε αλλά πάντως ήταν πολύ ζωφερός ο πίνακας που παρουσιάστηκε όχι τόσο ρόδινος όσο ακούγεται μερικές φορές στους δικούς σας κύκλους. και πρέπει πιστεύω να κάνουμε μια προσπάθεια εμείς ιδιαίτερως εκεί για να αντιμετωπιστούν τα, τα δυσάρεστα, τα αρνητικά στοιχεία στην ε, Τουρκία. Κράτησε περίπου μια μισή ώρα η συζήτηση. Όπως είπα, ό,τι σας είπα εδώ, ό,τι αρνητική εικόνα σας έδωσε εδώ για την κατάσταση στην Τουρκία, την μετέφερα και στον Πρωθυπουργό, ο οποίος με άκουσε με υπομονή Και πρέπει να πω προ το ζήτημα τη ασφάλεια. Βλέπουμε να έχουμε μια οπισθοδρόμηση στην κατάσταση που είχαμε πριν από τρία χρόνια περίπου, γιατί υπάρχει, φαίνεται, η ανάγκη για το κράτο να ενισχύσει τι συνθήκε ασφαλεία και να περιστείλει ω εκ τούτου τι ε, ελευθερίε ε, των πολιτών. Αυτό το ξεκίνησε οι ΗΠΑ μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Θεσπίστηκε αυτή η έννοια τη ασφάλεια, τη υπερκρατική θεωρία και τη ασφάλεια του κράτου και επεκτάθηκε και στα υπόλοιπε χώρε στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι ο μοναδικός ε, τρόπος, το μοναδικό μοντέλο για να ε, εξασφαλιστεί η ασφάλεια, η ηρεμία, η ειρήνη μέσα σε μια κοινωνία είναι οι ανθρώπινες ελευθερίες, είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διαφορετικά υπάρχει πάντα βία και μια κοινωνία που ζει μέσα στη βία δεν βρίσκει διέξοδο παρά μόνο με την προαγωγή των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Και πάλι μέσα στη διαδικασία του εκδημοκρατισμού λοιπόν, την οποία ε, να προχω... στην οποία απαιτείται να προχωρήσει η Τουρκία, πιστεύουμε, για τους λαούς μας, για τον τουρκικό και τον κουρδικό λαό, πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε στο βαθμό που μπορούμε. Τα ζητήματα της βίας δεν. Η, η βία δεν επιλύει προβλήματα. Αυτό το ε, επικαλούνται ακόμη και αυτοί οι οποίοι μετέρχονται βία στην ουσία. Για την ε, ερώτηση του φίλου μας για το αν το ΠΚΚ είναι τρομοκρατική οργάνωση, εγώ δεν έκανα ποτέ τέτοια δήλωση, γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη διαλεκτική μας από την αρχή, δηλαδή γιατί χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί βία, πού είχαμε φτάσει και χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί βία. Έτσι λοιπόν προτείνουμε να υπάρξει μια πρόταση, ένα μοντέλο, μια διατύπωση η οποία θα επιτρέπει την συμμετοχή μας ε, σε, μια, ε, σε ένα δημοκρατικό διάλογο. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλλουμε σε αυτόν ε, με όλες μας τις δυνάμεις. Είμαστε βέβαιοι ότι η κοινωνία απαιτεί αυτόν τον δημοκρατικό διάλογο για την ειρήνη. η στρατιωτική χούντα πολλές φορές ακούστηκε στην ομιλία μου γιατί θεωρώ ότι είναι υπεύθυνη υπέτεια για πολλά δυνά, διότι δεν υπήρξε κανένας μηχανισμός προστασίας της κοινωνίας από το κράτος. Ε, Ήταν σαν να έχει φτιαχτεί το κράτος για να προστατεύει τον εαυτό του και όχι τον άνθρωπο ή την κοινωνία. Και όμως το κράτος οφείλει να προσφέρει προστασία και ασφάλεια σε κάθε μέλος του, σε κάθε οντότητα που διαβιεί μέσα στα σύνορά του. Αυτά πιστεύω. Ευχαριστώ. Thank uh, um, Σας ευχαριστώ. Και για να σας ενημερώσω για τα θέματα των γυναικών και της ε, ισότητας των φίλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε 22 επιτροπές και μόνο 10 γυναίκες που είναι μέλη πρόεδροι αντιπρόεδροι, 34,8 είναι το ποσοστό των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 25% είναι γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 10 προεδρου επιτροπών που είναι γυναίκε έχουμε από 22 επίτροπε. Είμαστε κάτω από το 50% όπω βλέπετε. Έχω και μια επόμενη ομάδα ομιλητών. Θα ήθελα να σας ζητήσω να είσαστε σύντομοι στα ερωτήματά σας. Κυρία Κράτσα πρώτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, πιστεύω ότι είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για το κοινοβουλευτικέ επιτροπέ και τα μέλη του Κοινοβουλίου ευρύτερα η υποδοχή της κυρία Ζάνα, ε, βραβείο Ζαχάροφ του Κοινοβουλίου μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο εκτιμάμε την ανταλλαγή απόψεων μαζί σας και επίσης ήθελα να σας πω ότι η δημιουργία του δικτύου των βραβευμένων με το βραβείο Ζαχάροφ θα μας δώσει την ευκαιρία να έχουμε διάφορες εκδηλώσεις και ε, δυνατότητες να συνεχίσουμε το διάλογο, ε, να μαθαίνουμε το έργο σας και να εμπλουτιζόμαστε από αυτό, αλλά να σας δίνουμε και μια πλατφόρμα ε, συμβολής στην ανάγκη υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, σύμφωνα με την εμπειρία σας. Παρακολούθησα με ιδιαίτερη προσοχή την ομιλία σας και είδα ότι πέραν των κενών που υπάρχουν σήμερα στο κράτος δικαίου, στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, υπάρχουν και πενιχρές προοπτικές. Αυτό είναι το πολύ ανησυχητικό. Ήθελα να σας πω, σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών. Έχετε υπόψη σας την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση των γυναικών στην Τουρκία. Αν έχετε παρατηρήσεις να μας κάνετε από τη ζώσα εμπειρία σας, ή θα είναι πολύ χρήσιμη για μας, διότι θα την επαναλάβουμε αυτή την ε, προσπάθεια σύνταξη μιας έκθεσης την επόμενη χρονιά. Έχετε συναντήσει την εισηγήτριά μας, έχετε ανταλλάξει απόψεις μαζί της για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε κι εμείς ε, αυτές τις προκλήσεις μέσα στην έκθεση και στα ψηφίσματά μας. Είναι το πρώτο ερώτημά μου αυτό. Και δεύτερον, ε, μέσα στο κοινοβούλιο, μέσα στην οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, που έχει κάποια δομή ήδη στην Τουρκία, γίνεται συζήτηση για την ε, ε, ε, δυνατότητα αναβάθμισης των δικαιωμάτων των γυναικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ευρύτερα μέσα από την προσπάθεια της Τουρκίας για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετέχετε σε, κάποιους, σε κάποιες ομάδες συζήτησης προετοιμασίας του, ο, της προσαρμογής στο ευρωπαϊκό ε, κεκτημένο της Τουρκίας. Γίνεται σχετική συζήτηση στο Ευρωπαϊκ, στο, στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Εντάσσεται αυτούς τους προβληματισμούς στο διάλογο τον κοινοβουλευτικό στη χώρα σας για το πώς μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανταποκριθείτε σε αυτά τα, στις, αυτές μεγάλες προκλήσεις ε, ακόμη τις ε, προσπάθειες για δημοκρατία στην Τουρκία. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Madam Ευχαριστώ κυρία Κράτσα. Η κυρία Βεργιά έχει το λόγο. Κυρία Βεργιά. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς την Λέιλα Λάζανα και το θαυμασμό μου για το θάρρος και για την, ε, το μετριοπαθή τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τις απόψεις της μετά από αυτά τα οποία ζει, μετά από αυτά που έχει ζει στο παρελθόν, διατηρεί ακόμα την ίδια γαλήνη και νυφαλιότητα. Θα ήθελα να της θέσω μια σειρά ερωτήσεων υπομορφή τηλεγραφικών μονάχα κυρία Πρόεδρε. Παρουσιάσατε την κυρία Ζανά ως ανεξάρτητη βουλευτή. Θα ήθελα να μας εξηγήσει γιατί είναι ανεξάρτητη βουλευτής. Υπάρχουν πολλοί εκλεγμένοι στην αίθουσά μας. Γιατί είναι ε, ανεξάρτητη βουλευτής η κυρία Ζανά. Θα ήθελα επίσης να μας εξηγήσει για την ποια είναι η εξέλιξη της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας στην Τουρκία και πώς η Τουρκία έχει αυτό το λυπηρό προνόμιο να είναι η χώρα με τους περισσότερους κρατούμενους δημοσιογράφου στη φυλακή αυτή τη στιγμή. Το γεγονός επίσης ότι υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία δεν είχαν την τύχη να έχουν τη δυνατότητα να τύχουν μια δίκαιας δίκης. Ε, ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο χρησιμοποιείται η αντιτρομοκρατική νομοθεσία είναι πάρα πολύ σημαντική και θα, πρέπει, θα ήθελα να ξέρω και κάτι περισσότερο για τη δίκη των λεγόμενων κουρδικών κοινοτήτων, ΚΑΣΕΚΑ, γιατί μέσα στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας βρίσκονται οι περισσότεροι κρατούμενοι στη φυλακή αυτή τη στιγμή, βάσει της αντιτρομοκρατική ε, νομοθεσίας και τη υποτιθέμενης συμμετοχή του στο ΠΚΚ. Επίση, για τι βίες ενέργειε στην κουρδική πρωτοχρονιά, το Νευρός, και η βία η οποία έλαβε χώρα εφέτος κατά τη διάρκεια της, ε, του εορτασμού του Νευρός ήταν απόλυτα απαράδεκτη. Και επίσης αναφερθήκατε στις προσφυγές στο Συμβουλίο της Ευρώπης, στο ΕΔΑΔ. Εγώ υποστήριξα την απεργία πείνας στο Στρασβούργο και μία από, τις, ε, από τα αιτήματα των απεργών ήταν να αποσταλεί μια απο τις τα αιτηματα των απεργων ηταν να αποσταλει μια αντιπροσωπεια του Συμβουλίου της Ευρώπης από ό,τι γνωρίζω, η Επιτροπή ΣΕΠΕΤΕ, η Επιτροπή κατά των βασανιστήριων και της κακομεταχείρισης έστειλε μία αντιπροσωπεία, αλλά δεν μπόρεσε να πάει στην φυλακή όπου κρατείται ο κ. Σέτζαλάν. Θα ήθελα να μου επιβεβαιώσετε ή όχι αυτές τις ε, πληροφορίες. Και επίσης η δηλώση του κ. Σούλτς όταν γύρισε από την Τουρκία σε σχέση με την τελευταία καταδίκη που έγινε εναντίον σας ότι δεν ήταν δίκη αυτή η δίκη, ε, θα ήθελα να ξέρω τι θα έπρεπε να κάνουμε περαιτέρω για να σας υποστηρίξουμε ως βραβείο Σαχάροφ. Η κυρία Γκάμπριελ. Σας θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Ζάνα που είναι ανάμεσά μας σήμερα και θα ήθελα να ξέρετε κυρία μου ότι εντός αυτής της συνελεύσεως ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα, η προάσπιση του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αξιών της δημοκρατίας είναι στην πρώτη γραμμή και πάντα σας υποστηρίζουμε. Στην παρουσίασή σας, στην ομιλία σας εξηγήσατε τι πρέπει να γίνει και αυτό σε πολλά επίπεδα. Κυρίως υπογραμμίσατε την ανάγκη να δράσουμε εν πρώτης όσον αφορά την πολιτική βούληση και δέσμευση μακροπρόθεσμη. Είπατε όχι προσωρινά μέτρα. Λοιπόν, το πρώτο μου ερώτημα είναι, είμαστε παρουσία τέτοια πολιτική βούληση. Υπάρχει δέσμευση για την εξέβρεση μακροπρόθεσμη λύση για τι γυναίκε. Δεύτερον, υπογραμμίσατε σε θεσμικό επίπεδο ποιε είναι οι δυσκολίε. Αναφερθήκατε εκτενώ στα διάφορα κενά που υπάρχουν εντό του δικαστικού συστήματο όσον αφορά την αντιμετώπιση των διαφόρων υποθέσεων, καθυστέρηση των εκδικάσεων. Ερώτηση. Υπήρξαν ήδη ε, ποινές που ανακοινώθηκαν για, για βιοπραγίες κατά των γυναικών. Ξέρουμε ότι κάθε ένας που έχει υποστεί βία ε, για να μπορέσει να συνέλθει πρέπει να αισθανθεί ότι έχει δικαιωθεί. Και αυτό περνά το αίσθημα δικαιοσύνη μέσω ενό δικαστικού συστήματος που είναι αποτελεσματικότερο. Επίσης αναφερθήκατε στην ανάγκη να υπάρχει καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών εντός των θεσμών. Ε, το ερώτημά μου είναι απλό. Τι γίνεται Ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσει λήψεω πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων. Ε, ποια είναι τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν ούτω ώστε να βελτιωθούν τα δεδομένα. Ήδη αναφερθήκατε στο, στην επιθυμία σας να υπάρχει Υπουργείο Αρμόδιο για τις Γυναίκες. Εγώ θα ήμουν πιο διστακτική όσον αφορά αυτό. Πάντα φοβάμαι όσον αφορά τη δημιουργία ε, Υπουργείων για τις Γυναίκες. Μήπως δημιουργηθούν καταστάσεις ε, όπως στην Αφρική Οπότε αν δημιουργείται τέτοιο Υπουργείο ε, συμβάλλει στην ε, μείωση, στην καθυστέρηση των μαχών των γυναικών. Αντί να συνεχίσουν να πολεμούν και να δείξουν ότι τα, δικαιώματα των ανθρώπων, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δικαιώματα για τι γυναίκε, αυτό επέτρεψε η δημιουργία του Υπουργείου να στιγματιστεί κάπω η μάχη Στο τρίτο επίπεδο που αναφέρατε, τα ανθρώπινα δικαιώματα οι συνθήκε των γυναικών και των παιδιών στι φυλακέ για μία ακόμη φορά. Ποια μέτρα συγκεκριμένα θα μπορούσαν να ληφθούν για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση, ε, βράχη μέσω πρόθεσμα και όσον αφορά την πρόληψη των ε, βιοπραγιών, ε, τι μπορούμε να κάνουμε ε, πέρα από αυτά που ήδη επισημάνατε, πέρα από την επικύρωση του συμπληρωματικού πρωτοκόλου. κυρία Ζάνα, σας ευχαριστώ για τη διαδρομή που ακολουθήσατε. Επαναλαμβάνω την υποστήριξή μου και το πώς σας εκτιμώ. Σας ευχαριστώ. Thank you, ευχαριστώ κυρία Γκάμπρελ. Η Βαρόνι Λάτφορντ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ καλωσορίζω θερμά τη Λεϊλά Ζάνα. Χαίρομαι που την ξαναβλέπω. Έχει θάρρος τη μάχη που δίνει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κουρδικά δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτό το θάρρος είναι πολύ εντυπωσιακό και είναι χαρά να την βλέπουμε, όχι όμως χαρά να ακούω αυτά που έχει να μας πει. Νομίζω ότι μας παρουσιάσατε μια εικόνα σχετικά με τα διασυνδεόμενα ζητήματα. Ε, Έλλειψη ελευθερίας του κουρδικού λαού, ε, ε, οι επαγόρευση να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα τους, οι κρατήσεις χωρίς δίκη, φυλακής χωρίς δίκη, το ότι φυλακίζονται παιδιά και οι πολύ κακές συνθήκες στις φυλακές, όλα αυτά γνωρίζω ότι έχει παρακολουθήσει ποικιλοτρόπως ευσυρά ετών το Κοινοβούλιο. η πολύ ζωντανή παρουσίασή σας θα έπρεπε να μας αναγκάσει να συνεχίσουμε να ασχολούμεθα με όλα αυτά τα ζητήματα στο έργο μας. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω όμως, πιο συγκεκριμένα. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποιες λέξεις χρησιμοποίησατε, αλλά εξεπλάγει όταν είπατε νομίζω το εξής. η ενεργό συμμετοχή του Αμπτουλάχ Τσαλάν στην πολιτική συζήτηση και στην προσπάθεια εξέβρεσης πολιτικής λύσης του κουρδικού προβλήματος θα ήταν ευπρόσδεκτο από την κοινωνία της Τουρκίας, θα γινόταν αποδεκτό από την τουρκική κοινωνία. Εξεπλάγιν, διότι γνωρίζοντας το πώς εκείνος έχει δαιμονοποιηθεί για μεγάλο ποσοστό της κοινή γνώμης. Εκπλήσωμαι γι' αυτό. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε, να μου εξηγήσετε αυτή την παρατήρηση. Αν όντω έτσι έχουν τα πράγματα. Ανεξάρτητα τις απόψεις που έχει κάποιος για το ΠΚΚ και ότι θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση. Ο Τσαλάν σαφώς είναι ένα σύμβολο για τον κουρδικό λαό. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις συγκρούσαν και πρέπει να βρεθεί κάποια διέξοδος για πολιτικό διάλογο για να του δώσει κάποιο ρόλο. Και φαίνεται σαν να δίνεται κάποιες ελπίδες, Έχει, ότι υπάρχουν κάποιες ελπιδοφόρες προπτικές που δεν έχω ξανακούσει. Ευχαριστώ, Βαρόνι Λάτφορντ. Ο κύριος Ολμπιός, ο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι είμαστε εγωιτευμένοι από την παρουσία της Λεϊλάς εδώ σήμερα. Είναι μια μακρά ιστορία σχέσεων αλληλεγγύης μαζί της. Θα ήθελα όμως να προσθέσω ότι όλοι κατά πάσα πιθανότητα συμφωνούμε με τη γενική αυτή κατεύθυνση των πολιτικών αποφάσεων που δίνει η Λαζανά στην ε, συνάντησή μας. Γιατί η κατάσταση στην Τουρκία δεν είναι μια κατάσταση μονάχα που περιλαμβάνει πολύ σοβαρά προβλήματα, αλλά είναι μια κατάσταση μεγάλης πολυπλοκότητος και πολλών αντιμαχόμενων τάσεων για να καταλάβει κανείς αυτή την πολυπλοκότητα, η, η 24 Μαΐου καταδικάστηκε η κυρία ε, Ζλέιλα Ζανά σε 10 έτη φυλακής. Και στη συνέχεια, μετά από μερικές μέρες, βρίσκεται μαζί με τον ε, επικεφαλής της τουρκικής κυβέρνησης και συζητάει μαζί του. Νομίζω ότι το ερώτημα είναι για μένα, ήταν απλώς μια συμβολική και εφήμερη συνάντηση, μια πολιτική χειρονομία, είναι η απαρχή μιας πολιτικής η οποία θα μπορέσει να μας δώσει νέες ελπίδες. Είναι ένα στοιχείο λοιπόν το οποίο γεννά ελπίδες αυτή η συνάντησή σας με τον κύριο Ερντογάν, γιατί φυσικά ήταν αμφιλεγόμενη αυτή η συνάντηση, υπήρξαν πολλές απόψεις που διατυπώθηκαν σε σχέση με αυτή τη συνάντηση, σε σχέση με το περιεχόμενο αυτής της συνάντησης. Θα μπορούσατε να μας ε, βοηθήσετε να κατανοήσουμε καλύτερα αυτή την πολύπλοκη κατάσταση, λέγοντάς μας ποιες είναι οι τάσεις που αναδύονται σε σχέση με την ε, κουρδική και τουρκική πραγματικότητα και το αν βλέπουμε να υπάρχει κάποια απαρχή μιας διαδικασίας εγκατάλειψης της ένοπλης βίας και των στρατιωτικών επιχειρήσεων και της έναρξης ενός διαλόγου για την αναγνώριση των γλωσσικών και πολιτικών δικαιωμάτων του κουρδικού λαού. Ευχαριστώ, κύριε Ομπιόλς. Και εγώ έχω ένα σύντομο ερώτημα να θέσω. Περιγράψατε με μεγάλες λεπτομέρειες την κατάσταση στις φυλακές για τους πολιτικούς κρατουμένους και τους άλλους κρατουμένους. Μου φαίνεται βλέποντας ότι αυτή την κατάσταση ότι θα έπρεπε να επιληφθεί του θέματο αυτού ένα εθνικό θεσμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει περάσει πρόσφατα νομοθεσία στην Τουρκία για να δημιουργηθεί ένα θεσμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα μετά από μακρές και ουσιαστικές επικρίσεις των εθνικών και διεθνών μήκυο αυτής της νομοθεσίας. Υπάρχουν τώρα κάποιες βελτιώσεις και η Τουρκία έχει πλέον ένα νόμο προς την κατεύθυνση αυτή της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ποια είναι η άποψή σας για τη δημιουργία αυτού του φορέα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εθνικό επίπεδο στην Τουρκία. Και πριν σας δώσω το λόγο, είπατε στην αρχή, Λαϊλά Ζανά, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πράξει περισσότερα για να υποστηρίξει μια πολιτική λύση στην ε, σύγκρουση στην Τουρκία για την επίτευξη μιας διαδικασίας ειρήνευσης και θέλω να δώσω και στον εκπρόσωπο της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης το λόγο εν συντομία. Σας παρακαλώ να είστε πάρα πολύ σύντομος, γιατί ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει πολλά πράγματα για την Τουρκία σε διάφορα επίπεδα. Αν μπορείτε όμως να εστιάσετε αποκλειστικά μόνο σε ένα ή δύο θέματα και να είσαστε πολύ σύντομος. Και αν θέλει και η Λελάζα να μπορεί να σχολιάσει αυτό το θέμα. Down. Yes, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς κυρία Ντούμακ, δεν μπορεί να παρίσταται σήμερα. Θα διαβιβάσουμε το μήνυμά της γραπτός σε εσάς. Καλώς λέει η Πρόεδρος. Υπόσχομαι ότι θα ζητήσω γραπτή απάντηση που θα μπορέσω να προωθήσω μετά στη Λεϊλά Ζάνα ούτως ώστε να υπάρχει λεπτομερής ενημέρωση διότι γραπτός ε, υπάρχει όλος ο διαθέσιμος χρόνος και θα μπορεί να φανιστεί τι προετοιμάζεται λεπτομερώς. Από ό,τι είδα υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, υπήρχε κάποια λεπικάλυψη των ερωτήσεων, ίσως μπορείτε να ομαδοποιήσετε τις ερωτήσεις διότι έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας κατά 20 λεπτά, άρα πρέπει να είμαστε σύντομοι, έχετε το λόγο. tabii Πρέπει να επιμείνουμε ως προς τον μηχανισμό της δικαιοσύνης. Ο μηχανισμός λειτουργίας της δικαιοσύνης, εάν δεν υπάρχει σε μια κοινωνία, τότε είτε πρόκειται για τη σχέση μεταξύ ανδρών και γυναικών, είτε πρόκειται για τη σχέση μεταξύ των πολιτών και του κράτους, η κατάσταση συγχαίεται. Ε, ε, εμφανίζονται προβλήματα και μπερδέματα. Όταν έρχεται μπροστά τους ε, μια υπόθεση, οι δικαστές ε, μπορούν να την επεξεργαστούν μόνο με πολύ περίπλοκες διατυπώσεις, ε, μέσα από ένα βαρύ μηχανισμό, χρονοβόρο μηχανισμό και βλέπουμε ότι δεν δίνεται δικαιοσύνη. Είναι πολλοί αυτοί που έχουν κρατηθεί προσωρινά εν αναμονή μια δίκη και βρίσκονται χρόνια μέσα στι φυλακέ. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν αποδίδεται δικαιοσύνη, γιατί η δικαιοσύνη που καθυστερεί είναι μη δικαιοσύνη, είναι μη αποδοθήσα δικαιοσύνη. Σε αυτό λοιπόν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Ταυτόχρονα χρειάζεται μια προσπάθεια να αλλάξει η νοοτροπία προς τη συνημένη δικαιοσύνη. Το 1997 ήρθε από την Ελβετία να με επισκεφθεί στη φυλακή μια αντιπροσωπεία από την Ελβετία και με ρώτησαν τι πρέπει να κάνουν, τι μπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν. Ε, ε, η απάντησή μου ήταν ότι πρέπει εξάπαντος χωροφύλακες, αστυνομικοί και δικαστές να εκπαιδευτούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη δικαιοσύνη, σε θέματα δικαιοσύνης από την, ε, τις αρχές, τις ευρωπαϊκές κτλ. Έγινε μια προσπάθεια λοιπόν στην αρχή χωρίς πολλά αποτελέσματα. Πάντως μια μικρή αλλαγή είδαμε στην κοινωνία. Την περίοδο 99 με 2002-2003 υπήρξε μια μικρή πρόοδος. Οι αστυνομικοί δεν έπιαναν όποιο θέναν στον δρόμο να χτυπήσουν. Μπορούσε περπατάει ο δρόμος στους δρόμους ήσυχα. Ε, αλλά μετά, μετά δυστυχώ είδαμε μια οπισθοδρόμηση. Γύρισαν δηλαδή στα παλιά και οι αστυνομικοί και οι χωροφύλακε αλλά και οι δικαστέ. Άρα υπάρχει ζήτημα νοοτροπία. Άρα είναι ένα βαθύ πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα με πολλές ρίζες, ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει στη ρίζα του να αντιμετωπιστεί. Γιατί αν δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη, εάν ο δικαστής δεν αντιλαμβάνεται το πρόβλημα ως πρόβλημα ή το αντιλαμβάνεται αμερικώς, τότε δεν μπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν αρκεί η νομοθετική μερικώς, τοτε Πρέπει να αλλάξουν οτροπίες, πρέπει να αλλάξουν μυαλά Βεβαίω και χρειάζονται και νομοθετικέ ε, τροποποίησει και θεωρήσει αλλά και μάλιστα όχι με μικρά-μικρά βήματα. Πρέπει να αλλάξει ριζικά. Το Σύνταγμα, Φερρυπίν, ολόκληρο πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα το κρατικό. Εκεί που λέει δηλαδή το Σύνταγμά μα, μία είναι η γλώσσα, μία, ένα είναι το κράτο, όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν. Τώρα είμαστε στον 21ο αιώνα έχουν φτάσει οι κοινωνίε μα σε ένα επίπεδο στο οποίο δεν αρμόζει πλέον, δεν αντιστοιχεί πλέον και δεν ανταποκρίνεται στι ανάγκε του ένα τέτοιο σύστημα μονολυθικό. Είναι κάτι το οποίο συζητούμε, που πρέπει να συζητήσουμε, γιατί στην Τουρκία δεν έχει συζητηθεί ανοιχτά. Και το ζήτημα τη ε, ε, πρόθεση για μετάβαση σε ένα προεδρικό σύστημα. Πρέπει να συζητηθεί αυτό. Δεν μπορεί. Όπως αντίστοιχα και τα συστήματα, τα, το, το σύστημα που χρησιμοποιεί η Γερμανία, όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε. Δεν αντέχουμε πια άλλο, δηλαδή να συνεχίσουμε με ένα τέτοιο μονολυθικό βάρη σύστημα. Εμεί προσπαθούμε να συζητήσουμε τουλάχιστον το θέμα το προεδρικό. Έχει προξενήσει κάποιε συζητήσει. Θα είναι προεδρική, η προεδρευομένη όχι, ημιπροεδρικό το σύστημα. Όλα αυτά λοιπόν τα συζητούμε. Για τα παιδιά. Τα παιδιά δεν έπρεπε να είναι σε φυλακέ. Έπρεπε να είναι σε ε, κέντρα αναμορφώσεω ούτω πίν ε, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποδοθούν μετά στην κοινωνία. Δεν έπρεπε να είναι μέσα στις, ε, στα σοφρονιστήρια τα παιδιά. Και γιατί, γιατί πήρε μια πέτρα από το δρόμο να την πετάξει πάνω σε ένα τάγκ, πάνω σε ένα τεθωρακισμένο. Αυτό το παιδί πήγε φυλακή με τέτοια βαριά ποινή. Γιατί θεωρήθηκε επικίνδυνο για τις δομές του κράτους. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχθώ ούτε σαν άνθρωπος, ούτε σαν γυναίκα, ούτε σαν μάνα. Το ότι ένα τέτοιο παιδί πήγε φυλακή γιατί έπεσε μια πέτρα και τη σήκωσε απέναντι στο τεθωρακισμένο. Έπρεπε να είναι σε σχολείο, έπρεπε να είναι να μπορεί να φτιάξει τη ζωή του και να μορφωθεί. Για τον Οτζαλάν Νομίζω ότι θα πρέπει η κάθε κοινωνία να σκέφτεται και να αναλογίζεται τα δικά της, το δικό της συμφέρον, τη δική της ε, προτίμηση, να κάνει τη δική της επιλογή. Αυτό πρέπει να γίνει και στην Τουρκία. Εάν έχουμε τέτοια δυστημία, τέτοια ένταση στην Τουρκία αυτή τη στιγμή, εάν έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα ζωτική σημασία, εάν έχουν έρθει οι λαοί αντιμέτωποι ο ένας με τον άλλον, πρέπει να δούμε γιατί, πρέπει να δούμε γιατί μια τέτοια απόφαση έχει, έχει μια απόφαση περί ε, συζήτηση με τον Τσελάνο, ας πούμε, έχει τη δυνατότητα να προξενήσει δυσκολίες τόσο σοβαρές και να δώσουμε μια λύση. Πρέπει το ταχύτερο δυνατό δηλαδή να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό για να δοθεί λύση και τέλος στα προβλήματα. Πρέπει μια κοινωνία μόνη της να δίνει τα προβλήματα, στα προβλήματά της, ε, να μπορεί να μορφώνει τα παιδιά της, ε, να καθορίζει το μέλλον της, να μπορεί να διοχετεύει την οργή της, το, το, το, θυμό της. Και σε αυτό πιστεύω εγώ ότι δεν θα πρέπει η τουρκική κοινωνία να ε, αντιδράσει σε αυτό. Για δε την κουρδική κοινωνία μπορώ να σας πω ότι με κίνδυνο φυλάκισης, τιμωρίας, ποινών, κυρώσεων αναγνωρίζουν και εξακολουθούν να αναγνωρίζουν ως ηγέτη των Έχουμε 3,5 εκατομμύρια ποινέ, κυρώσει φυλακίσεις, ε, τουλάχιστον ε, δημόσιες, γιατί πώς, είναι, πώς έχουν υποστεί κυρώσει ε, κρυφέ και απόρριτε, δεν το γνωρίζουμε. Αλλά για αυτή την υπόθεση έχουμε πάρα, πολλές, πάρα πολλά δεινά υποστεί. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι δικαίωμα του κάθε λόγου και θα πρέπει ο καθένα μόνο να αποφασίζει. γιατί είμαι ανεξάρτητη βουλευτής. Να σας πω, αυτό είναι ένα άλλο μειονέκτημα του συστήματος Τουρκία. Μπορώ να εκλεγώ βουλευτής, αλλά δεν μπορώ να εκλεγώ ως μέλος κόμματος. Είναι λίγο παράξενο το, το γεγονός αυτό, η κατάσταση αυτή. Λοιπόν, όταν βγήκαμε από τη φυλακή το 2004 ως βουλευτές του Μπεντεπέ, τότε το, το, το είχε απαγορευτεί. Ιδρύσαμε λοιπόν το Μπεντεπέ, αλλά επειδή εμείς είχαμε απαγόρευση, είχαμε στέρηση πολιτικών ε, δικαιωμάτων, δεν μπορούσαμε να εκλεγούμε με το Μπεντεπέ. Μετά έκλεισε το Μπεντεπέ και σε ένα κογκρέσο εξελέγην εγώ ως εκπρόσωπος ε, μέλος της ε, συνέλευσης αυτή η εκλογή ήταν που θεωρήθηκε λόγος να απαγορευτεί το ΤΤΠ τότε. Είχα εκλεγεί εγώ από το λαό. Με έστειλε ο λαός στη Βουλή. Εγώ είμαι βουλευτής του Κοινοβουλίου, αλλά δεν μπορώ να είμαι μέλος του κόμματος που με έστειλε μέσω του λαού στην, ε, στη Βουλή. Άρα λοιπόν πρέπει αυτό το πράγμα να επιληθεί πλέον. Και όσο δεν αλλάζουν αυτά τα προβλήματα, όσο δεν καθαρίζει το πεδίο, δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουμε προς, ένα προς μια ουσιαστική αλλαγή στο Σύνταγμα. Ξέρετε ότι στην Επιτροπή που, που επεξεργάζεται το νέο Σύνταγμα υπάρχουν και βουλευτές του ΠΕΝΤΕΠΕ. Αλλά πρέπει να βρεθεί ένα κοινό πεδίο συνεννόηση, πρέπει να μπορέσουν... Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο ακόμα για να συνεχίσω. Έχω χρόνο καθόλου ακόμα, μπορείτε να μου πείτε αν έχω ένα χρονικό περιθώριο ακόμα να μιλήσω. Πέντε λεπτά, μάλιστα. Ευχαριστούμε. Πρέπει να ανοίξει το πεδίο λοιπόν. Να ανοίξει το πεδίο πρέπει να αντιμετωπιστεί το τουρκικό ποινικό σύστημα, το τουρκικό ποινικό κώδικα, το σύστημα ε, κράτηση στι φυλακέ, ε, το δικαίωμα υπεράσπιση του κρατουμένου, του κατηγορουμένου και όλα αυτά. Βεβαίω και το Σύνταγμα έχει τεράστια σημασία σε όλα αυτά, αποτελεί την απαρχή, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί και από την αλλαγή των νοοτροπιών. Η κοινωνία θα πρέπει να αποδεχθεί να απορροφήσει ούτω πίν ένα νέο σύνταγμα, ένα σύνταγμα δημοκρατικό, να το αποδεχθεί και να αλλάξει έτσι νοοτροπία. Αλλά εάν δεν μπορέσει ο πολίτης να έχει αρκετά δικαιώματα, εάν δεν υπάρχει γούρ ελευθερίες, δεν μπορεί οποιοδήποτε νέο σύνταγμα να φέρει ουσιαστική αλλαγή. Για την βία εις των γυναικών πρέπει να σας πω ότι αυτή ε, μπορεί να αντιμετωπιστεί ιδιαίτερα εάν η γυναίκα να λάβει δράση στον οικονομικό τομέα, στον οικονομικό βίο. Όταν δεν είναι παρούσα στον οικονομικό βίο η γυναίκα, είναι σαν ένας επέτης απέναντι στον άντρα της. Ένας ζητιάνος, με το χέρι απλωμένο. Γιατί, ούτε Γιατί και μετά από αυτό ούτε κοινωνική, ούτε πολιτική άνοδο μπορεί να περιμένει. Γιατί οικονομικά εξαρτάται από τον άντρα. Είναι επομένω σε θέση δευτερεύουσα, σε θέση αναπληρωματική, βοηθού δεν είναι εκείνη η οποία θα καθορίσει τις εξελίξεις και το μέλλον της. Και άρα στην πολιτική διαδικασία λήψη αποφάσεων πρέπει να αντιμετωπιστεί η γυναίκα ως άνθρωπος να μπορέσει η ίδια να διαμορφώσει το ε, μέλλον των γυναικών με βάση την γυναικεία θεώρηση. Πρέπει να είναι παρούσα η γυναίκα, πρέπει να βοηθήσει μία γυναίκα την άλλη, να προχωρήσει τη χειραφέτηση, να βοηθήσει μία την άλλη με την εκπαίδευση, με τη μόρφωση, με την παιδεία, έτσι ώστε η γυναίκα να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη περίοδο. Ξέρω ότι στην Ευρώπη υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία έχουν αντιμετωπιστεί ήδη από, τον, ε, από τα τέλη του 19ου αιώνα. Αλλά στην Τουρκία και ιδιαίτερα στο Κουρδιστάν όπου ε, είναι ξεχωριστή η κατάσταση, πρέπει η γυναίκα να κάνει ε, ακόμη πολλά βήματα, πρέπει να εξασφαλιστούν πολλά ακόμα βήματα για την ε, χειραφέτηση των γυναικών. Και ξέρετε βέβαια ότι αμέσως αντιδρούν οι άντρες, ανησυχούν γιατί θέλουν οι γυναίκες δικαιώματα, τι θέλουν να ζητήσουν, πού θα οδηγηθούμε κτλ. Πρέπει ω εκ τούτου να κάνουμε όλοι μαζί μια προσπάθεια. Η γυναίκα ως άνθρωπος ως γυναίκα, ως πολιτική δύναμη πρέπει να προχωρήσει. Αλλά για να προχωρήσει θα περάσει μόνο μέσα από την οικονομική χειραφέτηση. Με την οικονομική χειραφέτηση μπορεί κανείς να προσδιορίσει μόνο στο μέλλον του. Και γι' αυτό απαιτείται πάλι μόρφωση και παιδεία. Ξέρω ότι τέλειωσε ο χρόνος που είχα στη θέσή μου. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας απευθύνω τις θερμότερες ευχές μου σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή με την οποία με ακούσατε. Ίσως να μην έδωσα τις ε, ε, απαντήσεις σε κάθε ερώτηση σας διεξοδικά, αλλά όσο μου επέτρεπαν οι δυνατότητές μου, το έπραξα. Και προσπαθούμε πάντα, όπως είπα, να ε, προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι η ανάλυση σας, οι συστάσεις σας είναι, ήταν ιδιαίτερα καλόδεκτα στοιχεία εδώ και η Επιτροπή Γυναικών και η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο βαθμό του δυνατού προσπαθούμε να υποστηρίξουμε την ατζέντα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμάτων γυναικών στην Τουρκία και ιδίως στην περιοχή την Κουρδική. Ευχαριστώ. Okay, now I, we have really to be very quick πρέπει τώρα να βιαστούμε για να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημέρης της διάταξης για την κατάσταση των Ροχίνγκα στην Βυρμανία. Για αυτούς που πρέπει να φύγετε, παρακαλώ κάντε το γρήγορα. And, uh, uh, Σας υπενθυμίσω επίσης για αυτούς που παρακολουθούν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία στις 18 Σεπτεμβρίου θα εστιάσουμε στην κατάσταση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στα Δυτικά Βαλκάνια και στην Τουρκία. This is,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 Okay. Maybe you could just read the first two paragraphs of this one, leave out the rest, because she will explain anyway. So, now we have on our agenda the human... Έχουμε λοιπόν την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο κρατήδιο Ραχίνγκα στη Μιανμάρ. να κάνω μία εισαγωγή. Πόσο θετικές είναι οι εξελίξεις στο Μιανμάρ. Στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων το συζητήσαμε το θέμα πρόσφατα. Είχαμε και ψήφισμα τον Απρίλιο στο Κοινοβούλιο και έγιναν, διαπιστώσαμε τις βελτιώσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα που σημειώθηκαν. Σχεδόν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι απελευθερώθηκαν. Υπήρξε κατάπαυση του πυρός. Ε, υπάρχουν, ε, έγινε κατάπαυση του πυρός μεταξύ όλων των μειονοτήτων εκτός από μία και ελπίζουμε οι εξελίξεις να είναι θετικές. Ανησυχήσαμε για τα νέα που ακούσαμε, για την αύξηση των βίων επιθέσεων και συγκρούσεων ε, των μουσουλμανικών κοινοτήτων στο, τον Μάιο στο κρατήδιο Ραχίνε τον Μάιο και διερωτηθήκαμε χρειαζόταν ένα ψήφισμα στα κατεπήγοντα στο Κοινοβούλιο δεν κάναμε κάτι τέτοιο όμως και το συζητάμε τώρα στην Επιτροπή μας για να εξετάσουμε λοιπόν το θέμα αυτό, καλέσαμε τον, τον κύριο πρεσβευτή του Μιανμάρ και τον πρέσβη του Μπαγκλαντές. Δυστυχώς όμως είναι στη Νέα Υόρκη ο πρέσβης. Ευχαριστώ όμως που ήρθε άλλος εκπρόσωπος ε, της πρεσβείας του Μπαγκλαντές. Οι κανόνες της Επιτροπής μας προβλέπουν παρουσίαση του θέματος και αν ο πρεσβευτής εκπρόσωπος της πρεσβείας θέλει να πάρει το λόγο, μπορεί να το κάνει, αλλά θα πρέπει να περιοριστεί σε ένα τρίλεπτο. Συνολικά έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι τις 11 χρόνο για συζήτηση, αλλά έχουμε συγκεκριμένο θέμα για τους Ροχίνγκας, οπότε ε, μπορούμε να επικεντρώσουμε τη συζήτησή μας και τα συμπεράσματά μας. Καλέσαμε για παρουσίαση της καταστάσεως την κυρία Τιράνα Χασάν, που είναι ερευνήτρια της Human Rights Watch και στις 3 Ιουλίου επέστρεψε από την πρόσφατη αποστολή της Human Rights Watch στο Μιανμάρ όπου εξέτασε τη βία μεταξύ των εθνοτήτων, την όλη κατάσταση. Θα ήθελα να σας δώσω το λόγο τώρα για να μας ενημερώσετε για ένα πεντάλεπτο περίπου για την όλη κατάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομη γίνεται διότι δεν έχουμε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στη διάθεσή μας για να παρουσιάσουμε μια κατεπίγουσα και ενσυχητική κατάσταση. Ε, ήταν δύο εβδομάδες κράτηση η αποστολή μας για να εξετάσουμε τη βία στο Ρακάιν που είναι στη δυτική Βιρμανία. Ήταν σουρελιστική εμπειρία. Είχαμε τη βία λοιπόν που συγκλώνιζε τη δυτική Βυρμανία και χανόταν ανθρώπινες ζωές ενώ οι τηλεοράσει έδειχναν εικόνε της επίσκεψης τη Αξαουσί εδώ στην Ευρώπη. Και ήταν μια εποχή όπου ε, χαιρετίζονται οι μεταρρυθμίσει στη Βυρμανία και αυτό ήταν ε, μεγάλη αντίθεση με αυτά που βλέπαμε που συνέβαν στην Δυτική Βυρμανία αυτά που βλέπαμε και ακούγαμε τότε και θέλω να μοιραστώ μαζί σας λίγο αυτά που ακούγαμε αυτά που καταγράψαμε κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περίοδου αρχές Ιουνίου ε, υπήρχε βία μεταξύ εθνοτήτων μεταξύ της κοινότητας της μουσουλμανικής των Αχίγκα και των, των εθνοτικών βουδιστών Αρακάν Διάφορα επεισόδια οδήγησαν εκεί, αλλά στις 8 Ιουνίου στην πόλη Μοντόρ εκα, εκατοντάδες ε, ρίγκα ξεσηκώθηκαν, κατέστρεψαν διάφορα, διάφορους ναούς και σαν τύπηνα η Αρακάν σε κάποιες περιπτώσεις σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, την αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας βιοπράγησαν κατά των κοινοτήτων Ραχίνγκα. Δολοφονίες, ξυλοδαρμοί έκαψαν μουσουλμανικά χωριά και σπίτια. Η βία οδήγησε τεράστιες καταστροφές ε, περιουσιών, καταστάφησαν εκατοντάδες σπίτια. 90.000 ε, άνθρωποι εκτοπίστηκαν σύμφωνα υπολογισμού του ΟΗΕ. Επίσημο ο νεκρών ήταν 70 όταν κάναμε τι μετρήσει μα. Πιστεύουμε ότι είναι μεγάλη υποτίμηση του αριθμού των νεκρών. Είδαμε, είχαμε μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων που μας είπαν ότι 70 ε, άνθρωποι πέθαναν σε λίγες μέρες. Πολύ ε, μεγάλη βία και από τις δύο πλευρές, αυτό είναι κάτι που πρέπει να ερευνηθεί για τις βιοπραγίες, αυτό είναι αναμφισβήτητο, αλλά δυστυχώ σταμάτησε η καύση των χωριών, αλλά έγιναν άλλου είδους βιοπραγίες και καταχρήσεις που δεν σταμάτησαν. Νέο κύμα βιοπραγιών ξεκίνησε μετά από αυτές τις αρχικές συγκρούσεις και κατά κάποιο τρόπο χρησιμοποιήθηκε η αναταραχή αυτή ως, ε, ε, ε, ως, ως δικαιολογία για βιοπραγίες κατά τον Ραχίνγκα που είναι περιφερειακή. Οι μουσουλμάνοι Ραχίνγκα στη Βουρμανία θεωρούνται ως μη πολίτες. Αναφέρονται ως παράνομοι βεγγαλέζοι μετανάστες και δεν δέχονται ότι κατάγονται από τη Βερμανία ε, και δεν είναι αναγνωρισμένες μία από τις 135 αναγνωρισμένες εθνικότητες, δεν έχουν δικαίωμα ταυτότητας ε, πρέπει να καταγραφούν, να καταχω... έχουν προβλήματα για όσον αφορά τους γάμους, τις καταγνώριση γεννήσεων κλπ. Ε, και το καθεστώς το νομικό είναι πολύ αβέβαιο και γι' αυτό είναι ιδιαίτερα ευάλωτη όσον αφορά συστηματική παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίω στο βόρειο κρατήδιο του Ρακέιν. Λοιπόν, τι συμβαίνει στο βόρειο κρατήδιο του Ρακέιν. Πολύ δύσκολη η εικόνα, διότι η πρόσβαση σε αυτή την περιοχή είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Αλλά αυτό που κάναμε είναι μιλήσαμε με αυτόπτες μάρτυρες και επιβιώσαντες επιθέσεων και ίδιες ιστορίες ακούμε καθημερινά. Από όταν σταμάτησαν συγκρούσεις, οι δυνάμεις ασφαλείας που συμπεριλαμβάνονται τις περιφερειακές μεθοριακές αρχές, την ΑΣΑΚΑ, ε, αστυνομία, τους ΛΟΝΤΙΕΝ, την αστυνομία καταστολής ε, των ταραχών και στοιχεία του στρατού, όλοι αυτοί καθημερινά έκαναν σαρωτικές επιθέσεις και κατά τη διάρκεια αυτών των συλλήψεων των ε, ομαδικών εκατοντάδες συνελήφθησαν. Είναι με συνεχής διαδικασία φορτηγά φορτωμένα με νασάκα σάκα και δυνάμεις ασφαλείας φτάνουν σε ένα σχολείο και πόρτα με πόρτα κάνουν έρευνες, τραβάνε τον κόσμο από τα σπίτια τους, τους βγάζουν και τους δέρνουν. Οι Ραχίνγκα έχουν μακρά ιστορία ε, κα, ε, επιθέσεων από τους Νασάκα και όταν βλέπουν τους Νασάκα να φτάνουν στο χωριό τους κάνουν ό,τι θα έκανε οπισδήποτε από μας. Τρέχουν, το βάζουν στα πόδια. Και όπως τρέχουν τους πυροβολούν. Τους πυροβολούν με, με, με, πυκνά πύρα. Και αυτοί που είναι αρκετά τυχεροί να μπορέσουν να διασχίσουν τον ποταμό, να κολυμπήσουν, να το σκάσουν και να τρέξουν αρκετά γρήγορα, βλέπουν τα δέντρα και βλέπουν τους θείους τους, τα αδέρφια τους, τις θείες τους, τα παιδιά τους να πυροβολούνται. Μερικοί από αυτούς σκοτώνονται, κάποιοι αφήνονται εκεί τραυματισμένοι. Για εκείνους που δεν μπορούν να διασχίσουν, να τρέξουν αρκετά γρήγορα, αυτοί καταδιώκονται, τους καταδιώκουν οι δυνάμεις ασφαλείας, τους κυνηγάνε, τους σταματάνε, τους δέρνουν, τους δένουν, τους έχουν επιτεθεί με σπαθιά, τους έχουν πυροβολήσει, τους έχουν δύρει και τους ηλικιωμένου και τα παιδιά και αυτό δεν είναι κάτι που συνέβη επειδή υπήρξαν συγκρούσεις τώρα Ρακάν. Είναι κάτι που είδαμε να συμβαίνει την περασμένη εβδομάδα και το καταγράψαμε. Στις έρευνές μας λοιπόν Καταγράψαμε διάφορες παραβιάσεις, αλλά επειδή δεν έχω πολύ χρόνο θα προχωρήσω ε, και θα αναφερθώ σε αυτά που πρέπει πραγματικά να γίνουν. Συστηματικά υπάρχουν αυτές οι παραβιάσεις, είναι φρικαλές οι πράξεις που διαπράττουν οι δυνάμεις ασφαλείας. Είναι πήγον, κατεπήγον, διεθνή αυτιά και μάτια να είναι επιτόπου στο Ρακάιν. Ε, την περασμένη εβδομάδα όταν ε, κάναμε τις έρευνές μας εκεί ακούσαμε ότι ένα ψήφισμα θα πέρναγε από το Κοινοβούλιο, θα εγκρινόταν από το Κοινοβούλιο και λυπηθήκαμε πάρα πολύ όταν δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Αλλά υπάρχει ακόμα χρόνος, γνωρίζω ότι όλοι πάτε για στερινές σας διακοπές σύντομα αλλά σας παρακαλώ, σας παρατρύνω, χρησιμοποιήστε αυτό το διαθέσιμο χρόνο για να δραστηριοποιηθείτε διότι οι παραβιάσεις που μιλάμε, αυτές οι πράξεις ε, γίνονται σήμερα. Και Ερκούλες, σε σχεδία σχεδόν, ε, προσπαθούν να πιαστούν και στο από ένα πλαστικό δοχείο για να κολυμπήσουν, να περάσουν το ποτάμι για να μπουν στον Μπαγκλαντές. Και όταν τα καταφέρνουν να μπουν στον Μπαγκλαντές, δεν υπάρχει προστασία εκεί πέρα. Δεν τους ε, αναγνωρίζει το καθεστώς του πρόσφυγα τους ξαναβάζουν στις παλιόβαρκες και τους ξαναστέλνουν πίσω μέσα από τις βροχές ε, του Μουσόνα ε, και πιστεύω στην κατάσταση που σας ε, περιέγραψα. Σας παρακαλώ λοιπόν, κάντε ένα-δύο μικρά πραγματάκια στο χρόνο που έχει σε θέση σας και θα ήθελα να σας παρακαλέσω, σας εκλυπαρώ, είναι κατεπήγον εκατοντάδες άνθρωποι μπαίνουν σε κρατήσεις χωρίς καμία επικοινωνία από τον έξω κόσμο, τους συλλαμβάνουν και εξαφανίζονται. Χθε το βράδυ συνέβη αυτό, προχθές συνέβη, απόψε μπορεί να συμβεί αυτό. Λοιπόν, θα σας ενεθάρρυνα να προσπαθήσετε να διεξαχθεί μια ανεξάρτητη έρευνα. Να μπορέσετε εσείς να υποστηρίξετε τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για τη Βυρμανία και τις διάφορες αποστολές που γίνονται εκεί να διαθέσετε πόρους ούτως ώστε να υπάρξει ανεξάρτητη έρευνα. Η κυβέρνηση συμφώνησε ότι θα πρέπει να διεξαχθεί μια έρευνα, αλλά η Επιτροπή Έρευνας που προτάθηκε αποτελείται από μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που πραγματοποιούν αυτά τα πράγματα που σας περιέγραψα. Αυτό δεν είναι ικανοποιητικό. Πρέπει να γίνει πλήρης ανεξάρτητη έρευνα. Δεν υπάρχει χρόνος, αλλά δεν είναι αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο. Τι πρώτε εβδομάδε του Ιουνίου περάσαμε χαιρετίζοντα μεταρρυθμίσει ενώ η Άγκ Σουνσί ήταν εδώ και επισκεφτόταν την Ευρώπη. Ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό, μεν, αλλά δεν είναι αυτό που χρειάζεται για να λάβει χώρα μεταρρύθμιση. Για να γίνει πραγματική μεταρρύθμιση πρέπει να υπάρξει λογοδοσία για σοβαρές φρικαλαιότητες κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτή είναι η δοκιμή που πρέπει να γίνει. Το νέο πακέτο για τα ανθρώπινα δικαιώματα καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τις παραβίασεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να τους δικάσει. Να είστε όσο αυστηροί όσο με το Σουδάν, όσο με τη Συρία, όπως με το Μαλί. Έτσι παρομοίως να προσεγγίσετε και τις δράσεις σας σχετικά με τη Βυρμανία. Ευχαριστώ κυρία Χασάν που μας δώσατε μια, από, το πρώτο χέρι πληροφόρηση. συντομία δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο Τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να μας πει τι γίνεται σε αυτόν τον τομέα από αυτή την υπηρεσία. Ε, thank Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν ζωφερή η εικόνα που παρουσιάστηκε στην, για τη Βερμανία. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αυτές τις πληροφορίες, σίγουρα όμως θα τις εξετάσουμε. Η δική μας εικόνα της κατάστασης επιτοπίως είναι ότι τα πράγματα έχουν γαλινέψει σε κάποιο βαθμό, ότι οι εντάσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων παραμένουν φυσικά. Υπάρχει ο κίνδυνος αναζωπήρωσης των ε, πράξεων βίας. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν εκτοπιστεί 90.000 άτομα, 10.000 βουδιστές Ρακίνοι και 80.000 μουσουλμάνοι που βρίσκονται σε προσωρινούς καταβλισμούς και σε μοναστήρια αυτή τη στιγμή. Κατανοούμε ότι η κυβέρνηση δίνει έκτακτη ανακουφιστική βοήθεια, τρόφιμα, στέγαση και έκτακτη βοήθεια υγειονομική. Ζητά διεθνή βοήθεια. Η πρόσβαση από διεθνείς ΜΚΟ και από, το, από τα Ηνωμένα Έθνη έχει επιτευχθεί σε κάποιο βαθμό, αλλά λόγια ασφαλείας εμποδίζουν την πλήρη ανάπτυξη αυτών των ε, ενεργειών Ξέρουμε ότι 10 μέλη των ιατρών χωρίς σύνορα και της υπάτης ε, αρμοστίας για τους πρόσφυγες είναι αυτή τη στιγμή υποκράτηση, χωρίς να έχει απαγγελθεί καμιά κατηγορία. Γνωρίζουμε επίσης και πρέπει να το λάβουμε το υπόψη ότι υπάρχει η διαδεδομένη αντίληψη ότι η διεθνής αρρωγή έχει ευνοήσει δυσανάλογα το μουσουλμανικό πληθυσμό και λόγω των βιαίων γεγονότων αυτό μεταφράζεται σε μια αρνητική και εχθρική στάση προς τις ξένες υπηρεσίες και μικιό και το προσωπικό τους. Όλα αυτά τα θέματα τα θίξαμε χθες το πρωί με τους ε, υπεύθυνους με τον υπεύθυνο υπουργό, τον υπουργό για τα συνοριακά θέματα και μας είπανε ότι ο ίδιος ο πρόεδρος επέμεινε ενώπιον του επικεφαλής του δικαστικού τομέα ότι πρέπει να ακολουθηθεί η σωστή διαδικασία σε δικαστικό επίπεδο και για τους συλληφθέντες από τις οργανώσεις βοήθειας και όλα αυτά χωρίς καμία πολιτική παρέμβαση. Το Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συμμετάσχει σε μια επίσκεψη επιτοπίως για να αξιολογήσουν την κατάσταση και οι συνάδελφοί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να σας δώσουν περισσότερα στοιχεία. Πρέπει να σας πω επίσης ότι μετά από το 2001 η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους κύριους παρόχους υποστήριξης στην περιοχή του, στην επαρχία Ρακίν. Καλύπτουμε θέματα όπως είναι ε, έργα αποχέτευσης, ε, εξυγίανσης, ε, εκπαίδευση κτλ. Εξακολουθεί όμω να υπάρχει η υπόνοια και η κατηγορία εναντίον μα ότι είμαστε μεροληπτικοί στι παρεμβάσει μα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρος. Και ο Ασκόν, την, ε, ο επικεφαλής της, ε, του τμήματος για τις ε, δράσεις είναι παρόν. Σας παρακαλώ, αν θέλετε να λάβετε λόγο, να είσαστε σύντομος. επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Απλώς να συνδέσω αυτά που είπε, που, με αυτά που είπε ο συνάδελφος από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Το ΕΚΟ, το Γραφείο Ανθρωπιστικής ε, Βοήθειας, βρίσκεται στην Μιανμάρ εδώ και πολλά χρόνια ως δωρητής. Η αρρωγή μας, το μεγαλύτερο μέρος της έχει πάει στην πολιτεία του Ραχίνε. Έχουμε λοιπόν δώσει υποστήριξη και στην ομάδα αυτή των ε, Ραχίνγκα και μας ανησυχούν τα μάλα τα πρόσφατα γεγονότα τα οποία καταδεικνύουν και πάλι την ανάγκη να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα σε πιο μακροχρόνια βάση. Αλλά αυτό που μας αφορά άμεσα είναι τα πρόσφατα γεγονότα και αυτό που επιζητούμε είναι να, είναι να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί που έχουν ανάγκες, αυτοί που έχουν εκτοπιστεί, ήταν τα θύματα της βίας, όλοι αυτοί που έχουν επηρεαστεί από τα γεγονότα αυτά, ότι είναι απαραίτητο όλοι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν την απαραίτητη βασική βοήθεια που χρειάζονται. Οι εταίροι μας που εργάζονται στην ε, πολιτεία του Ραχάν είναι έτοιμοι να βοηθήσουν. Το ΕΚΟ είναι έτοιμο να δώσει την απαραίτητη χρηματοδότηση. Η πρόκληση όμως που αντιμετωπίζουμε τώρα μαζί με τους εταίρους μας είναι ότι η πρόσβαση στην περιοχή αυτή έχει περιοριστεί σημαντικά λόγω της έκρηξης βίας. Δεν είναι μονάχα το θέμα του να πάρει κανεί την άδεια να μεταβεί στην περιοχή αυτή, αλλά υπάρχει και ένα κλίμα εχθρότητας εναντίον των ανθρωπιστικών οργανώσεων, εναντίον της διεθνούς κοινότητος, το οποίο είναι ιδιαίτερα ανισχυτικό και δυσκολεύει ιδιαίτερα τους εταίρους μας στην παροχή βοήθειας. Θέλουμε να παροτρύνουμε λοιπόν τις αρχές της Μιανμάρ να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό με έναν τρόπο ο οποίος θα κάνει δυνατό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια η οποία πρέπει να παραδοθεί κατεπηγόντως. Υπάρχει τώρα περιορισμένη πρόσβαση όπως σας είπα, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα, ιδίω για τις πιο απομεμακρυσμένες περιοχές, για τις οποίες δεν έχουμε πληροφορία τι γίνεται. Έχουν γίνει λοιπόν κάποιες εκτιμήσεις για τις ανάγκες σε επίπεδο ε, επισητισμού υπάρχουν προβλήματα, υπάρχει υποσιτισμός σε πολλές περιοχές, αλλά δεν μπορούν να δράσουν οι εταίροι μας λόγω της κατάστασης ασφαλείας και της έλλειψης πρόσβασης. Ένα άλλο θέμα το οποίο θέλω να σας αναφέρω είναι το γεγονός ότι κάποια από τα μέλη του προσωπικού της υπάτης αρμοστίας για τους πρόσφυγες και τους εταίρους τους είναι ακόμα υποκράτηση. Η Επίτροπος μας, η κυρία Γεώργεβα, που ήταν στην Ιαπωνία την προηγούμενη εβδομάδα για μια διάσκεψη, είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Υπουργό Εξωτερικών της Μιανμάρ και έθιξε το θέμα αυτό, το θέμα της πρόσβασης, <clears throat> αλλά επίση και ζήτησε και μια εξήγηση από τις αρχές της Μιανμάρ για την αυθαίρετη κράτηση ενός αριθμού εργαζομένων στις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Κάτι ακόμα για τον Μπαγκλαντές. Δεν έχουμε πληροφορίες για άφηξη νέων κυμάτων ε, τον άσυλο από την πλευρά της Μιανμάρ στο Μπαγκλαντές. Αυτό όμως το οποίο θέλω να πω σήμερα είναι το εξής, ότι και από την πλευρά του Μπαγκλαντές γίνεται δύσκολη η ανθρωπιστική πρόσβαση οι λίγοι εταίροι που έχουμε εκεί και οι οποίοι εργάζονται με χρηματοδότηση της ΕΚΟ για να βοηθήσουν περίπου 30.000 ε, μη νόμιμους μετανάστες από την ε, περιοχή του Ραχίνε στον Μπαγκλαντές έχουν μεγάλες δυσκολίες να φέρουν σε πέρα στο έργο τους και ζητάμε από την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να τους δώσει τις απαραίτητες διευκολύνσεις. Είμαστε σχεδόν η μόνη χορηγή στην περιοχή αυτή. <clears throat> Αν θα πρέπει να φύγουν αυτές οι οργανώσεις που υποστηρίζουν τους μετανάστες από τη βάση τους όπου λειτουργούν, τότε οι μετανάστες αυτοί θα μείνουν χωρίς καμία υποστήριξη και αυτό θα έχει δραματικές συνέπειες σε ανθρωπιστικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Και ρωτώ αν θέλει κανείς άλλος να λάβει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Τανκία τον ε, πρεσβευτή για την παρουσία του εδώ και τον ακούμε. Σα Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και θα προσπαθήσω να περιορίσω στα τρία λεπτά που μας έχετε δώσει. Η κατάσταση αυτή προκύπτει μετά από κάποια επεισόδια στα τέλη Μαΐου το βιασμό την ε, και τη ληστεία εις βάρος βουδιστριών γυναικών και μετά βίες επιθέσεις που οδήγησαν στο φόνο 10 μουσουλμάνων της Μιανμάρ μέσα σε ένα λεωφορείο. Έτσι λοιπόν άρχισαν στάσεις σε τρεις ε, κομοπόλεις με 77 νεκρούς, με δεκάδες ε, χιλιάδων σπιτιών, ε, και πολλών μοναστηριών και άλλων εγκαταστάσεων που ε, παραδόθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν. Στις 11 Ιουνίου απευθυνθεί έκκληση για συνεργασία των Αναστασιαστών με την κυβέρνηση για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου. Η κυβέρνηση έχει θεσπίσει 89 ε, στρατόπεδα υποδοχής των αστέγων μετά τις ε, στάσεις, της περιοχές αυτές και καλεί τις θρησκευτικέ οργανώσεις, τα πολιτικά κόμματα, τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών και τους προύχοντες των κοινωνιών να συνεργαστούν. Ήταν ε, πρωτοβουλίε αυτέ που χαρακτηρίστηκαν ευπρόσδεκτε από την διεθνή κοινότητα. Ο δε κύριο Φιτζινάμπιερ, ειδικό ε, σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στη συνέχεια επεσκέφθη το κρατήδιο Νάμπτζετ, μίλησε με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη Στη συνέχεια επισκέφθηκε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου μας ε, τα στρατόπεδα αυτά υποδοχή των αστέχων, συζήτησε με τις τοπικές αρχές ε, για, την, ε, για τα μέτρα ε, αντιμετώπισης των προβλημάτων, για την αποκατα... προσπάθεια και αποκατάσταση του κράτους δικαίου. Έγιναν επίσης επισκέψεις στις 2 Ιουλίου συγκεκριμένα έγινε μια επισκέψη στο Μπαγκλαντές για την αμοιβαία συνεννόηση πανστροπό αντιμετώπισης των προβλημάτων με, με ένα μνημόνιο που γράφηκε για την αμοιβαία συνεννόηση στα θέματα αυτά. Η Μιανμάρ, κυρία Πρόεδρε, είναι μια από τις πιο πολύχρωμες, πολύμορφες χώρες της περιοχής. Έχουμε πολλούς διαφορετικούς πληθυσμούς που συνεπάρχουν στη χώρα αυτή εδώ και αιώνες. Αυτές οι στάσεις πάντως έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και αποτελούν οπισθοδρόμοι σε σχέση με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για αναθεώρηση της κυβέρνησης, για ε, μεταρρυθμίσεις της κυβερνήσεως. Ε, επιδεινώνεται το πρόβλημα των ε, μεταναστών επίσης και πρέπει να γίνουν ε, προσπάθειες για τη μετώπιση αυτών των προβλημάτων, για την επούλωση αυτών των πληγών και για την εξασφάλιση ηρεμίας και τάξης έχει ξεκινήσει το Κοινοβούλιο και το, ο νομοθέτης θα αναθεωρήσει και θα μεταρρυθμίσει νομοθεσία που χρειάζεται να τροποποιηθεί ε, συμπεριλαμβανομένων και διατάξεων του συντάγματος αν χρειάζεται για τις εθνωτικές ομάδες. Αυτό που θέλουμε είναι η, ο λαός της Μιαμάρ, όλοι οι κάτοικοι στη Μιαμάρ να έχουν ε, τις ίδιες δυνατότητες για συνύπαρξη, δυναμική συμβίωση, για ανάπτυξη και ε, ζωή μέσα σε ένα δημοκρατικό και ειρηνικό έθνος. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη και τώρα στρέφομαι προς, την, προς τον εκπρόσωπο της Πρεσβείας, ο, ο εκπρόσωπος του Μπαγκλαντές, ο κ. Τσασταφέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Εκ μέρους της Πρεσβείας θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ενδιαφέρον της για αυτό το θέμα. Σχετικά με αυτό θα ήθελαμε να αναφέρουμε ότι η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές παρακολούθησε τις εξελίξεις στην πολιτεία αυτή του Μιανμάρ και θλίβει για την απώλεια ζωών και των περιουσιών λόγω των βιοπραγιών. Ελπίζουμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα ζητήματα θα αντιμετωπιστούν με το σωστό τρόπο και ότι η ειρήνη και η σταθερότητα τελικά θα επικρατήσουν στο ΡΑΚΕΝ. Το Μπαγκλατές δεν είναι μέρος της συμβάσεως του 1950 της πρόσφυγες, ούτε στο πρωτόκολλο του 67 αλλά δεν έχουν παρόλα αυτά αρνηθεί προστασία, ε, στέγαση και υποστήριξη στους Ραχίνγκα ε, για λόγους κατεπήγους ανθρωπιστικής ανάγκης. Πρόσφατα οι Ραχίνγκα του Μιανμάρ που προσπάθησαν να μπουν στον Μπαγκλατές εθράφησαν, τους δώσαν φάρμακα και καυσίμα για τους κινητήρες των σκαφών τους και τους ε, δώσαμε κίνητα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Ελπίζουμε ότι συμφιλωτικό ρόλο τη κυβερνήσεω του Μιανμάρ και των διαφόρων δυνάμεων τη τάξη θα αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη μεταξύ του, των Ραχίνγκα, ούτω ώστε να επιστρέψουν Ραχίνγκα. Σχετικά με αυτό, θα θέλαμε να πούμε κάτι που ανέφερε και ο προσευχή του Μιανμάρ. Πρόσφατα έγινε διαβουλεύση του Υπουργείου Εξωτερικών. Συζητήσει Μπαγκλαντέ και Μιανμάρ στην Τάκα και επανέλαβε ο, ο υφυπουργό του, ε, του Μιανμάρ ότι, θα δεχτούμε τους πρόσφυγες στο ε, Ελπίζουμε να επιστρέψουν τελικά όμως στην πατρίδα τους χωρίς καθυστέρηση και με αξιοπρέπεια να μπορέσουν να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Νομίζω ότι ακούσαμε τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς και ελπίζω ότι διάφορες δραστηριότητες ΕΚΟ, υπηρεσίες εσωτερικής δράσης και του ΟΗΕ που γίνονται επιτόπου και, από και στην πλευρά του Μιανμάρ και στην πλευρά του Μπαγκλαντές να συνεχιστούν αυτές οι δράσεις και να βελτιωθεί η διάδραση αυτών των ενεργειών με τους ε, επισήμους φορείς του Μπαγκλαντές και του Μιανμάρ ούτως ώστε να υπάρξει άμεση βοήθεια ε, να σταματήσει ε, το πρόβλημα και να βοηθηθούν οι άνθρωποι εκεί. Μακροπρόθεσμα είναι πολύ περίπλοκο το ζήτημα και κύριε Πεσβευτά είπατε ότι το Κοινοβούλιο συνεδριάζει τώρα. Ε, νομίζω είναι κάποιο που είναι μέλος του Κοινοβουλίου, τουλάχιστον αν επισκεφθήκαμε το Μιανμάρ, που είναι από την κοινότητα των Ροχίνγκα και θα μιλήσει για αυτό το θέμα. Και μακροπρόθεσμα ο καθένας που ζει στο Μιανμάρ έχει το δικαίωμα έχει το δικαίωμα του να έχει μια ηθαγένεια. Και ίσως μακροπρόθεσμα αυτό θα πρέπει να εξεταστεί. Διότι αν κάποιος έχει την ηθαγένεια, την υπηκότητα, εκείνος ή εκείνοι έχουν και δικαιώματα που του αρμόζουν. Κυρία Χασάν, είπατε ότι έρχονται οι θερινές διακοπές για το Κοινοβούλιο αλλά στεφόμενοι που συναδέλφους μου λέγω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα, ότι θα σταματήσουμε στο να σκεφτόμαστε και να, ότι, δεν θα, ότι δεν θα καταλήξουμε ε, σε κάποια συμπεράσματα να αποστείλουμε και στο Ban moon ε, και να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη και αυτά που κάνει η ΕΚΟ Επιτόπου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους που ήρθατε εδώ και που συζητήσαμε αυτό το θέμα, το οποίο είναι πραγματικά κάτι φοβερό για τον κόσμο εκεί. Σας ευχαριστώ να σας πω ότι μεταρρυθμιζόμαστε σε μια κεκλεισμένων ε, των θυρών συνεδρίαση τώρα του διευρυμένου Προεδρίου.